Liebe Kolleginnen und Kollegen. συνεχίζεται η συνεδρία της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και περνάμε στο σημείο 6 της διάταξης ανταλλαγή απόψεων και πληροφοριών με την Επιτροπή Εποπτείας της Αρχής Καταπολέμησης των Απατών, Όλαφ. Η ανταλλαγή αυτή απόψεων είναι κάτι το τακτικό. Ως Επιτροπή Ελέγχου έχουμε συχνά τέτοιες συνεδριάσεις. Όμως αυτή η συγκεκριμένη ανταλλαγή απόψεων γίνεται σε μια πολύ ιδιαίτερη συγκυρία. Καταρχάς καλωσορίζω τον κύριο Ντένολφ καθώς και την κυρία Σόμπρη και την κυρία Πινιόν, καθώς και τους κυρίους Μπέρς και Τίμεμανς. Τους καλωσορίζω θερμά όλους αυτούς. Όλη λοιπόν η, εποπτική, η Επιτροπή Εποπτείας είναι παρούσα, χαίρομαι ιδιαίτερα γι' αυτό. Η συνεδρίες είναι δημόσια, οπότε δύο λόγια ε, για την συγκυρία λοιπόν για να είμαστε όλοι απόλυτα ενήμερη Δεν είναι καθημερινό ένα μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να έχει ε, δηλώσει ότι θα παραιτηθεί. Και καθόλου συνηθισμένο δεν είναι μετά την ε, παρέτησή του να κυκλοφορούν διάφορες ε, φήμες για το εάν ήταν θελούσια ή όχι η παρέτηση αυτή δεν θα πω τίποτα γι' αυτό, αλλά η Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού θεωρεί ότι εφόσον είναι αρμόδια για την καταπολέμηση των απατών, για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, θα ήθελε σε μία μη δημόσια συνεδρίαση των συντονιστών να συζητήσει με τον Τζοβάνι ε, Κέσλα, επικεφαλής που είναι αρμόδιος για την υπηρεσία αυτή για να έχουμε την ευκαιρία να μας παρουσιάσει την άποψή του. Ο κύριος Κέσλερ το έκανε αυτό. Και στο τέλος αυτής της κεκλεισμένα των θυρών ανταλλαγής απόψεων τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου και ο αρμόδιος της Όλαφ κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι θα ήταν σκόπιμο να κάνουν τις εξής συστάσεις προς τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου. Πρώτον, να επιτρέψουν στα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου του Προπολογισμού ε, να έχουν πρόσβαση στα κείμενα για τη σχετική ε, υπόθεση και επίσης ε, να προτείνουν στον κύριο Μπαρόσο να λάβει θέση επί της παρέτησης του Επιτρόπου Ντάλι το Προεδρείο συμφώνησε και ο κύριος Σούλτς έστειλε μια επιστολή στον πρόεδρο Μπαρόζο. Λάβαμε την απάντηση του κυρίου Μπαρόζο και θα διανεμηθεί στα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ώστε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασής μας είτε στη συνεδρία των συντονιστών να συζητήσουμε αυτή την απάντηση. Κατά τη γνώμη μου είναι πολύ λογικό εφόσον παρετείται ένας επίτροπος, να έχουν τη δυνατότητα τα εκλεγμένα μέλη του Κοινοβουλίου να συζητήσουν με τον πρόεδρο τη Επιτροπής τους λόγους που οδήγησαν σε αυτή την παρέτηση. Επειδή λοιπόν είναι αυτό το πολιτικό πλαίσιο, δεν είναι εύκολο να συζητήσουμε με εσά τώρα για τα γενικά καθήκοντα της Επιτροπής Εποπτείας, οπότε να τονίσω ότι επειδή ε, είναι σημαντική και η συζήτηση για το νομοθετικό καθεστώς του Όλαφ, της Όλαφ, σκόπιμο λοιπόν είναι που δημιουργήθηκε η, Όλα, η Όλαφ και είναι οπωσδήποτε αναγκαίο να έχει τις αναγκαίες θεσμικές ρυθμίσεις για να καταπολεμήσει τις απάτες. Το 1990 δημιουργήθηκε η Όλαφ, τονίστηκε τότε η ανάγκη ανεξαρτησίας αυτής της αρχής, το τονίζω αυτό, για το Κοινοβούλιο πάντα ήταν σημαντική αυτή η ανεξαρτησία. Εφόσον όμως είμαστε ένα δημοκρατικό καθεστώς, λόγω του διαχωρισμού των εξουσιών και του δημοκρατικού ελέγχου, ένα τέτοιο ανεξάρτητο σώμα πρέπει να υπόκειται στο δημοκρατικό έλεγχο με βάση την αρχή των ελέγχων και ισορροπιών. Η εποπτική λοιπόν ε, αρχή, η Επιτροπή Εποπτείας της Όλαφ έχει ένα πολύ σημαντικό ρόλο να παίξει. Χαιρόμαστε λοιπόν πολύ που είναι παρόντες εδώ οι εκπρόσωποι της Επιτροπής Εποπτείας της Όλαφ και θα θέλαμε να ακούσουμε την άποψή σας για το τι σας απασχολεί αυτή τη στιγμή, πόσο θεωρείτε ότι είναι αποτελεσματική η εργασία σας και τι αναμένεται από εμά ω υποστήριξη του Κοινοβουλίου πώς μπορούμε όλοι να συνεργαστούμε για να εφαρμόσουμε τον καλύτερο τρόπο την ε, νομοθεσία της Ένωσης. Αυτά ω εισαγωγή και να δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Ντένολφ, επικεφαλή της Επιτροπής Εποπτεία. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Τόερ. Καταρχά να ευχαριστήσω την Επιτροπή Ενέχου Προπολογισμού που δέχτηκε το αίτημα για τη σημερινή συνεδρίαση. Η κυρία Κάστερ πήγε στην Εποπτική Επιτροπή πριν τον Απρίλιο. Από αυτή την επίσκεψη πολλά συνέβησαν εκ των υστέρων. Επιμείναμε να συναντηθούμε τον Κοκομπίου διότι ανήκει σε τα θεσμικά όργανα που μας διόρισε. Πριν συναντήσουμε τους εκπροσώπους της Βουλής των Λόρδων που μας κάλεσαν να συζητήσουμε μαζί τους την λειτουργία, την ελεγκτική της Υποπτικής Επιτροπής. Η Εποπτική Επιτροπή Τη Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης απάτη, δημιουργήθηκε για να ενισχύσει την ανεξαρτησία τη Όλαφ μέσω τακτικής παρακολούθησης των ερευνητικών λειτουργιών αυτής συγκρατούμενη από το να παρεμβαίνει ε, στην διεξαγωγή των ε, ερευνών. Η Επιτροπή ε, ελέγχει κατά πόσο διεξάγονται σωστά έρευνε τη Όλαφ. Η Υποπτική Επιτροπή βοηθά και τον Γενικό Διευθυντή τη Όλαφ στην απαλλαγή του, στην αντιμετώπιση των ευθυνών του. Στόχος της Επιτροπής είναι να υποστηρίξει το έργο της Όλαφ και να φροντίσει ούτως ώστε το ερευνητικό της έργο να διεξάγεται σύμφωνα με τις υψηλότερες προδιαγραφές εν πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών. Απαλλάς, δίνεται απαλλαγή μέσω υποβολής εκθέσεως στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και χορηγώντας γνωμοδοτήσεις στο Γενικό Διευθυντή υποβάλλοντας ερωτήσεις, συστάσεις ε, για την Όλαφ για βελτιώσεις όταν αυτό θεωρείται ως κάτι ενδεδειγμένο και αναγκαίων. Η Εποπτική Επιτροπή ενεργά και τακτικά παρακολουθεί τον τρόπο με τον οποίο διεξάγονται οι έρευνες από πλευράς ε, Όλαφ. Μόνο μέσω συνεχών προσπαθειών εξετάζοντας αντιπροσωπικό δείγμα διαφόρων υποθέσεων και συζητώντας υποθέσεις με τους, ερευνη... τους αρμόδιους της Όλαφ είναι δυνατόν να εντοπιστούν εάν υπάρχουν πιέσεις επί της Όλαφ που υπονομεύουν την ανεξαρτησία της. Και τώρα η Εποπτική Επιτροπή έρχεται στην Κοκομπύ κατόπιν δική της πρωτοβουλίας, ούτω ώστε να εξηγήσει τα προβλήματα που αντιμετώπισε στην εκπλήρωση της αποστολής της. Ήτι τον τακτικό, τακτική παρακολούθηση της εφαρμογής των ερευνητικών λειτουργιών της Όλαφ. Ο Γενικός Διευθυντής δεν συμφωνεί με το βαθμό των νομικών εξουσιών που διαθέτει η Εποπτική Επιτροπή. Από την αρχή της χορηγής εντολής, η Εποπτική Επιτροπή αντιμετώπισε προβλήματα όσον αφορά την πρόσβαση σε στοιχεία υποθέσεων όπου έπρεπε να κάνει τον έλεγχο των ερευνών της Όλαφ, η δική μας Επιτροπή. Ο Γενικός Διευθυντής της Όλαφ καθυστέρησε ή και αρνήθηκε την πρόσβαση σε φακέλους επικαλούμενους ε, κανόνες ε, προστασίας των δεδομένων. Γι' αυτό η Επιτροπή μετά από μακρές συζητήσεις με τον Γενικό Διευθυντή συμφώνησε ότι θα, ε, θα πρέπει, θα, λειτουργούσε τα πέσα του Solvit για την προστασία των δεδομένων. Και το 2007 όμως αυτό καλύφθηκε από σχετική γνωμοδότηση αν κινούμεθα εντός των ορίων. Παραθέτω, έτσι περαιτέρω, μια μεθοδολογία θα καταρτιστεί που θα περιγράφει τα διάφορα βήματα που θα πρέπει να ακολουθούνται σε οποιαδήποτε αίτημα πριν από την πρόσβαση σε όλους τους φακέλους CMS. Στο τελευταίο βήμα, το τελευταίο βήμα, η εποπτική αρχή αποφασίζει κατά πόσο τα πρώτερα βήματα υπήρξαν ανεπαρκή για την επίτευξη του ρόλου τους, για την ε, υλοποίηση του ρόλου και, και αν χρειάζεται πρόσβαση στον πλήρη φάκελο. Η Όλαφ θα πρέπει να σημειώσει στο σύστημα που διαχειρίζεται τους φακέλους ε, κατά πόσον ε, μπορεί να εγκρίνει την πρόσβαση της Εποπτικής ε, Επιτροπής. Αυτό σημαίνει ότι η Όλαφ δεν έχει δικαίωμα να αρνηθεί όμως πρόσβαση. Και επίσης δεν προβλέπεται η αδίποτε καθυστέρηση όσον αφορά τη χορήγηση αδείας για την πρόσβαση στους φακέλους. Σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες που διέπουν τη λειτουργία τη Οπτική Αρχή Επιτροπής και σύμφωνα με τις ρυθμίσει που συμφωνήθηκαν με τον Γενικό Διευθυντή της Όλαφ, η Επιτροπή θα πρέπει να λαμβάνει τις κατάλληλε πληροφορίε για υποθέσει που διαβιβάζονται στι εθνικέ δικαστικέ αρχέ τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν από τη σχετική διαβίβαση. Υποχρέωση πρώτερης ενημέρωσης πριν τη διαβίβαση απορρέει από το άρθρο 11.7 της αποφάσεως 1093 του 99 ως ερμηνεύτηκε από το Γενικό Δικαστήριο και διάφορες υποθέσεις, αποφάσεις που ελήφθησαν ούτω ώστε να ελέγχει κατά πόσο προστατεύονται τα θεμελιώδη δικαιώματα. Η Επιτροπή μα να ελέγχει κατά πόσο γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι βασικέ αρχέ όταν γίνεται έρευνα για κάποιο άτομο. Όμω διόρισε η Επιτροπή τον εισηγητή από την στιγμή που εγκρίθηκε η πρόσβαση στου σχετικού φακέλους. Η εξέταση τη σωστή διεξαγωγή τη έρευνα έχει ξεκινήσει. Αυτή η εξέταση πρόκειται να ολοκληρωθεί σύντομα και η Επιτροπή στην επόμενη ολομέλειά της θα αποφασίσει για τα επόμενα δέοντα βήματα. Αυτή η τελευταία παράγραφος αφορά η υπόθεση η οποία είναι πολύ ανοιχτή και αναφέρεται στο διεθνή τύπο. Η Εποπτική Επιτροπή της Όλαφ, κατά την άποψή μας, είναι κρίσιμος θεσμός που παρακολουθεί τη διενέργεια των ερευνών από πλευράς Όλαφ λόγω της πλήρους αυτονομίας και ανεξαρτησίας του Γενικού Διευθυντού της Όλαφ σχετικά με αυτό το θέμα. Η Εποπτική Επιτροπή πράγματι είναι ο μόνος φορέας που παρακολουθεί τις έρευνες της Όλαφ και νομίζω ότι είναι σημαντικότατο αυτό να το υπενθυμίζουμε. Η, ερευνητική αυτή επιτροπή για να λειτουργεί σωστά, η Εποπτική Επιτροπή, ε, πρέπει να πληρούνται οι κάτωθοι συνθήκες. Πρώτη, πρόσβαση στις υποθέσεις, στους φακέλους, όποτε η Επιτροπή θεωρεί κάτι τέτοιο αναγκαίο. Κάτι που έχει επιβεβαιωθεί από το ε, EDPS όπως προανέφερα, από το σύστημα επεξεργασία των φακέλων. Δεύτερον, θα πρέπει να σέβεται όλου του κανόνε η Όλαφ και τους κανον, τον εσωτερικό κανονισμό τη Επιτροπής που ε, έχει δημοσιευθεί στην επίσημη εφημερίδα. Τρίτον, ανεξάρτητη λειτουργία και σωστά στελεχωμένη γραμματεία τη Επιτροπή. Αυτή η ανεξαρτησία δεν είναι εγγυημένη αν μπορεί να αλλάζει ο Γενικό Διευθύνσης όλα το προσωπικό καταβούληση. Και το έκανε αυτό ε, από 8 άτομα έγινε το προσωπικό 6. Πλήρης έλεγχος της Επιτροπής του προπολογισμού της, συμπεριλαμβανομένων όλων των δαπανών της Γραμματείας, που σημαίνει ξεχωριστό κονδύλι του προπολογισμού. Ζητούμε να μας βοηθήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να πληρούνται αυτοί οι όροι, να γίνονται σεβαστοί οι προαναφερθέντες όροι, αυτό ήταν επίσημο σημείωμα της Εποπτικής Επιτροπής που προετοιμάσαμε και ήταν σημαντικό να το γνωρίζετε αυτό ότι αυτός και μόνο αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο παριστάμεθα εμείς εδώ σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Ντενόλθ, για τη δήλωση αυτή εκ μέρους της Εποπτικής Επιτροπής και θα δώσω το λόγο στα μέλη της Επιτροπής. Η ε, κυρία Κρέστρε είναι η πρώτη. Ευχαριστώ. Ω εισηγήτρια για την νομική βάση της Όλαφ, χαίρομαι πολύ που ήρθατε σήμερα και σας ευχαριστώ. Αυτά που μας τα είπατε δημόσια τα συζητήσαμε πριν και, και κλεισμένων των θυρών. Και νομίζω ότι είναι εντελώ απαράδεκτο αυτό που έκανε ο Γενικός Διευθυντής που πρέπει να ελέγχεται από εσά. Και έχουμε προσπαθήσει πολύ για να σας ε, ε, αναδείξουμε και να σας δώσουμε και δυνατότητες εργασίας. Δεν μπορεί ο Γενικός Διευθυντής της Όλαφ να περιορίζει τις δυνατότητες εργασίας σας. Δεν θα το δεχτεί αυτό η ομάδα μου άλλο. Καθίσαμε επί ένα χρόνο και παρακολουθούσαμε πώς παρεμποδίζεται η δουλειά σας και παλιά ό,τι είχε συζητηθεί δεν τηρήθηκε Μέχρι τώρα δεν υπήρχε Επιτροπή Εποπτείας, αλλά δεν θα το δεχτούμε πια άλλο αυτό. Ε, έχουμε χάσει πάρα πολύ χρόνο και ε, αν δούμε και τις λεπτές αποχρώσεις της υπόθεσης Ντάλι, νομίζω ότι πρέπει να ενδυναμώσουμε και όχι να αποδυναμώσουμε ε, το καθεστώς. Για το, την επόμενη χρονιά έχουμε κάνει μια πρόταση και προσπαθούμε να περάσει αυτή η γραμμή του προϋπολογισμού και επίσης ε, και προσπαθούμε να επιβάλλουμε και το σωστό οργανόγραμμα για την Επιτροπή Εποπτείας, αλλά το πρόβλημα είναι βαθύτερο. Γιατί όταν ο Γενικός Διευθυντής ε, δεν δέχεται τους διαδικαστικούς κανόνες, ε, αυτούς που έχετε δεχτεί και από τους προκατόχους σας, δεν τους φτιάξατε εσείς, οι κανόνες αυτοί ανέκαθεν ίσχυαν. Πώς είναι δυνατόν ξαφνικά να μην ισχύουν επειδή αυτός που πρόκειται να ελεγχθεί θέλει να αποφαίνεται επί των κανόνων του ελέγχου και του τρόπου του ελέγχου. Εάν δεν αντιδράσουμε θα κάνουμε ένα τεράστιο λάθος. Λοιπόν, ε, ε, το γάντι αυτό της πρόκλησης εγώ θα το σηκώσω. Ο, η, η Κομισιόν και ο Επίτροπος Σέμετα που κάθεται και κοιτάει πώς ε, εσείς στριμώχνεστε με την πλάτη στον τοίχο δεν είναι σωστό. Ε, εγώ δεν θα τον δεχτώ πια. Θέλω να κάνετε τη δουλειά σας, να μπορείτε να έχετε πρόσβαση και στο σύστημα διαχείρισης των υποθέσεων χωρίς να ε, παρεμβαίνετε στις τρέχουσες ε, εργασίες, δεν είναι αυτό η δουλειά σας άλλωστε. Πρέπει λοιπόν να κάνετε τη δουλειά σας και ο Γενικός Διευθυντής δεν σας αφήνει. Δεν είναι δική μου, δεν τα βγάζω από το μυαλό μου αυτά, εσείς τα είπατε. Είναι εντελώ απαράδεκτο αυτό που συμβαίνει αφού μάλιστα εσείς πρέπει να τηρείτε το σεβασμό στους κανόνες. Λοιπόν, θα πρέπει να, εφόσον αυτοί οι κανόνες δεν γίνονται σεβαστοί, θα πρέπει να αναζητήσουμε να δούμε και άλλους που έχουν τυχόν παραβιαστεί. Και επειδή είναι, ε, τρέχει διαδικασία ντάλι, ε, δεν ξέρω, ίσως θα έπρεπε να σας καλέσουμε πάλι και όταν θα έρθετε στην Επιτροπή θα μας υποβάλλετε έκθεση ό,τι μπορείτε να μας πείτε. Επίσης θα με ενδιέφερε να μου πείτε την ε, έκθεση, την Olaf Report, πότε τη λάβατε, με ποια ημερομηνία. Με ενδιαφέρει επίσης η εκτίμησή σας σχετικά με, την, ε, το συμβατό, με την απόφαση Φρανσέ Μπικ που λέει στην παράγραφο 164 ψάχνω αλλά δεν τη βρίσκω. Η παράγραφος ε, το 164 λέει, για την ερμηνεία δηλαδή του 1073 κανονισμού και λέει ότι η έρευνα αυτή έγινε πριν από την, ε, πρέπει να γίνει πριν από, τις από την ε, απασχόληση των δικαστικών αρχών. Είπαμε ότι το άρθρο 13.5 στον κανονισμό πρέπει να εφαρμοστεί δηλαδή γιατί ο χειρισμό του θέματος. Ε, είναι πολύ σημαντικό για μένα να μου πείτε τη γνώμη σας, ε, πώς θα γίνει δηλαδή, πώς θα ασχοληθούν πριν αποσταλεί στα κράτη-μέλη στη Μάλτα η υπόθεση Ντάλι, γιατί η περίπτωση Ντάλι προφανώς ε, μας ταρακουνάει όλους σχετικά με το τι επιτρέπεται και τι δεν επιτρέπεται. Αυτό είναι το διακύβευμα στην υπόθεση Ντάλι ευχαριστώ πολύ. Είναι κεντρική σημασία στο θέμα αυτό. Και εγώ θα προσθέσω αμέσως άλλη μια ερώτηση. Σε αυτά τα πλαίσια έγιναν ανακοινοθέντα τύπου για την αλλαγή στην Προεδρία της ε, Επιτροπής ε, Εποπτείας. Ε, και μια και είστε εδώ μπορείτε να επιβεβαιώσετε αυτές τις δηλώσεις του τύπου, στον τύπο. Δηλαδή διαδικαστικά μπορείτε να μας πείτε τι έγινε και τι διδάγματα, αν θέλετε, πρέπει να αντλήσουμε από αυτά όλα. Γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις, και το είπατε, οι προθεσμίες που περιλαμβάνονται και στη νομική βάση πρέπει να τηρηθούν. Έπαιξε αυτό, δεν έπαιξε αυτό κεντρικό ρόλο. Ευχαριστώ πολύ για τις δύο ερωτήσεις. Εάν, από ό,τι κατάλαβα τουλάχιστον, η πρώτη ερώτηση. Υπόθεση Φράνσι Μπέκ, την απόφαση. Είπαμε ότι ο Γενικός Διευθυντής της Όλαφ δεν συμφωνεί με το δικό μας εσωτερικό κανονισμό. Σε όλους τους εσωτερικούς κανονισμούς αναφέρεται ότι εάν πληροφορηθούμε από την Όλαφ περί μίας υποθέσεως θα πρέπει να διορίσουμε εισηγητή. Το κάναμε αυτό. Ότι πρέπει να περιμένουμε για την έκθεση του εισηγητού να υποβληθεί αυτή στην επόμενη ολομέλεια της αρχής εποπτείας, της Επιτροπής Εποπτείας και εξ αυτού δεν μπορούμε να αποκαλύψουμε τίποτα πριν συζητηθεί στην ολομέλειά μας που προβλεπόταν 22, μάλλον προβλέπεται 22 Νοεμβρίου. Σε αυτή τη φάση είμαστε τώρα. Δηλαδή, στο στάδιο που βάσει του εσωτερικού μας κανονισμού διορίσαμε εισηγητή, ετοιμάζει η εισηγήτρια την έκθεσή της, η κυρία Πινιού είναι η εισηγήτρια, ετοιμάζει την έκθεσή της που δεν είχε τη δυνατότητα να την υποβάλει ακόμα στην ολομέλειά μας. Δεν είμαστε υπάλληλοι πλήρους απασχόλησης, αλλά συναντώμεθα τακτικά, μια φορά το μήνα. Περιμένουμε να υποβληθεί η έκθεση πριν αυτό, εάν σεβαστούμε το δικό μας εσωτερικό κανονισμό, δεν μπορούμε να το κάνουμε. Εμείς σεβόμαστε τον εσωτερικό κανονισμό, δεν τον σέβεται ο Γενικός Διευθυντής τη Όλαφ. Τώρα για την παρέτηση του πρώην Προέδρου της Επιτροπής Εποπτείας. Το συζητήσαμε και κλεισμένο των θυρών. Και είμαι σίγουρος ότι και το Κοινοβούλιο διεξάγει συζητήσεις και κλεισμένων των θυρών και το σεβόσαστε αυτό. Κάναμε, ετοιμάσαμε ανακοινωθέν τύπου επίσημο. Και εγώ παραμένω σε αυτή τη θέση. αυτού, αυτή είναι η θέση μου, αυτή είναι η απάντησή μου. Όλοι έχουν το δικαίωμα να συζητούν και κλεισμένων των θυρών και νομίζω, αν έχω δίκιο, ότι τα θεσμικά όργανα να αποκαλύπτουν τα όσα συζητήθηκαν ε, και κλεισμένων των θυρών είναι και κάτι κολάσιμο. Ευχαριστώ. Βεβαίως ε, σεβόμαστε αυτό που δεν συζητείτε δημοσία. Αλλά επειδή αυτά τα θέματα συζητούνται δημοσία, καλό είναι να δίνετε εδώ η δυνατότητα να μας ενημερώνετε. Και ο κύριος ε, Τίμερμανς θέλει κάτι να πει. Ορίστε. Ευχαριστώ, πολύ, Πρόεδρε. Uh, ε, διάβασα και εγώ στον τύπο, ιδιαίτερα το γερμανικό, πολλά πράγματα για τους ε, λόγους της παρέτησής μου ως Προέδρου. Αυτή η πληροφόρηση είναι εντελώς αστήρικτη και πραγματικά με σοκάρισαν αυτές οι δηλώσεις και οι αναφορές στον τύπο. Εμείς ως Επιτροπή Εποπτείας υποβάλαμε ένα ανακοινοθέν στον τύπο που έλεγε εγώ, ότι εγώ παρατήθηκα από πρόεδρος για προσωπικούς λόγους. Προτιμώ να τους κρατήσω προσωπικούς τους λόγους αυτούς. Παρακαλώ. Δεν είμαι έτοιμος να συζητήσω το θέμα αυτό. Ελπίζω να είναι κατανοητό και να είναι και σεβαστό. Ευχαριστώ. Η συνάδελφος, ο συνάδελφος Ινσκάγε. Ich habe äh, dich zuerst Εσένα είδα πρώτο. Σίγουρα πρέπει να την κάνουμε κάποια στιγμή αυτή την κουβέντα με ενδιαφέρει όμως να κάνουμε σωστές διαφοροποιήσεις, να ξεχωρίζουμε τα πράγματα. Έχουμε συνάντηση, είχαμε συνάντηση για κλεισμένο των θυρών με τον ε, Διευθυντή Κέσλερ στο Στρασβούργο και θέλω να ερμηνεύσω το αποτέλεσμα. Μια ομάδα βουλευτών θεωρούν τον Ντάλι αθώο, άλλοι πάλι βουλευτές θεωρούν ότι ο Ντάλι είναι ένοχος. Κανείς βέβαια δεν αποφάσισε πάνω σε συγκεκριμένη βάση. Μόνο από τις εφημερίδες έμαθαν ότι έγινε έρευνα της Όλαφ που δόθηκε στις αρχές της Μάλτας και τώρα, και μάλλον όχι, δεν, δεν υπάρχει σαφής κατηγορία που λέει ότι είναι ένοχος, ε, αλλά η υπάρχουν κάποιοι που λένε θα δούμε τι θα κάνουν και οι αρχές της Μάλτας. Από την άλλη πλευρά έχουμε πειθαρχική ε, διαδικασία από την Κομισιόν. Οι άλλοι έλεγαν ότι κάτι ε, ε έχει κάνει, κάτι, υπάρχει που βρήκε η Όλαφ. Δεν ξέρουμε ποιος έχει δίκιο και αν ο Ντάλι με βάση τις ε, κατηγορίες ε, του δικαίου της Μάλτας ε, είναι ένοχος ή όχι, αυτό δεν έχει αποφασιστεί. Εγώ είπα στη συνάντηση των συντονιστών ότι δεν μπορώ να κρίνω. Γιατί πάνω σε ποια βάση θα κρίνω την υπόθεση αυτή. Μόνο από τον τύπο έμαθα και την συνάντηση με τον κύριο Κέσλερ, ο οποίος απάντησε και όπως και άλλοι συνάδελφοι απάντησαν και το μόνο που μπορώ να πω είναι το αν ο κύριος Μπαρόζο έδρασε στα πλαίσια του πειθαρχικής διαδικασίας ε, σωστά ή όχι. Πάνω σε αυτή τη βάση υποστήριξα την ιδέα που παρουσίασε ο πρόεδρος Θόιρερα ότι θέλουμε παρακαλώ πολύ να ξέρουμε την έρευνα της Όλαφ. Είπα και στους συντονιστές βέβαια ότι αυτό μπορεί να μην μας βοηθήσει, γιατί αν ξέρω εκ των υστέρων Δηλαδή δεν ξέρω στοιχεία και πώς να αξιολογήσω ε, τη θέση του εισαγγελέα ή και των άλλων παραγόντων. Ε, θα πρέπει να δούμε και τις συνθήκες πλαίσιο της Όλαφ και τις συνθήκες πλαίσιο για την ολοκλήρωση της, της έρευνας. και από εκεί θα πρέπει να κάνω κάποια αξιολόγηση εγώ ως Ευρωβουλευτής. Τώρα συζητάμε δύο πράγματα, έτσι κατάλαβα εγώ. Το ένα είναι μπορεί η Επιτροπή Εποπτείας της Όλαφ να δουλέψει σωστά. Γιατί είδα ότι υπάρχουν κάποιες ενστάσεις, ότι κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει. Αυτό είμαι πρόθυμος να το συζητήσω, γιατί η Επιτροπή Εποπτείας της Όλαφ έχει συγκεκριμένη λειτουργία, η οποία είναι προσδιορισμένη και αν οι συνάδελφοι από την Επιτροπή Εποπτείας της Όλαφ θεωρούν ότι δεν ε, υπάρχουν σωστές συνθήκες για τη δουλειά τους, αυτό πρέπει να το λάβω υπόψη μου. Αλλά δεν μπορεί να τα ανακατεύουμε αυτά με την υπόθεση Ντάλι, γιατί έτσι μπερδεύονται τα πράγματα και συζητάμε για μια δεύτερη διάσταση ξαφνικά που δεν τη γνωρίζομαι επί της ουσίας τόσο καλά. Εκτός ε, και αν πρόκειται για θέματα ε, που, αφορά, που έθεσε η ε, Ίγκε. Πότε δόθηκε η έκθεση στις αρχές της Μάλτας. Λοιπόν, στον κανονισμό λέει shall inform, δηλαδή ο Γενικός Διευθυντής θα ενημερώσει, το έκανε, διενημερώνει. Πρέπει να ενημερώσει πριν από την παράδοση στις αρχές της Μάλτας, το έκανε. Τώρα το αν είναι ε, σωστό το διάστημα των πέντε ημερών και όχι το διάστημα των τριών ημερών, να το δούμε. Αλλά νομίζω ότι τα, κατάκανε αυτά. Γι' αυτό θα συνεβούλευα παρακαλώ να αφήσουμε απ' έξω την υπόθεση Ντάλι το τι έγινε θα μας το πει η Επιτροπή Εποπτείας μετά την ολοκλήρωση των διαβουλεύσεων που δεν έχει γίνει ακόμα και όλα τα άλλα μένουν όπως ήταν και την προηγούμενη εβδομάδα. Το αν, κάποιο, ο, άνθρωπος ε, παρέπεσε σε σφάλμα θα το διαπιστώσει η ποινική διαδικασία, η ποινική δίωξη, γι' αυτό διορθώνω δεν ήθελα να χρησιμοποιήσω τη λέξη ένοχος στην αρχή και δεύτερον, το αν ήταν πειθαρχικά σωστή η διαδικασία, αυτό ευχαρίστως να το συζητήσω με τον κύριο Μπαρόζο, κανένα πρόβλημα. Αλλά τώρα θα πρέπει να δούμε πού είναι τα προβλήματα, ε, ε, ποια είναι τα προβλήματα με τον κύριο Κέσλερ, τι ε, πόρους διαθέτεται, σας τους πήραν πίσω, με ποια νομική βάση θα κάνετε καταγγελία εναντίον του. Αυτά είναι που θέλω να συζητήσουμε σήμερα το απόγευμα μαζί. Και την υπόθεση Ντάλι παρακαλώ ας την αφήσουμε κατά μέρος. Ευχαριστώ πολύ κύριε Γκάιερ. Ο συνάδελφος Μούλντερ. Δύο θέματα τίθενται εδώ. Πρώτα, έχουμε κανονισμό. Και σε αυτόν περιγράφεται το καθήκον της Εποπτικής Επιτροπής. Ακούω ότι η Εποπτική Επιτροπή δεν είναι απόλυτα ικανοποιημένη με τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να λειτουργήσει. Αυτό δεν είναι θέμα ατομικό δύο ατόμων, αλλά της ίδιας της Όλαφ και της εποπτικής αρχής. Θα το καλωσόριζα αν ο διευθυντής της Όλαφ ήταν εδώ παρόν, ούτω ώστε έτσι άμεσα να μπορούσε να τοποθετηθεί επί των οικασιών που ακούστηκαν σήμερα από πλευράς της Εποπτικής Επιτροπής. Ακούσα μόνο τη μία πλευρά. Θα πρέπει, θα πρέπει να ακούσουμε και από τις δύο πλευρές. Γιατί ο διευθυντής της Όλαφ δεν σας δίνει το περιθώριο να κινηθείτε όπως θεωρείτε ότι θα έπρεπε. Αυτό θα ήταν κάτι που θα ήθελα να γνωρίζω. Για την υπόθεση Ντάλι. Σαν κοινοβούλιο κάναμε αυτό που έπρεπε από τη στιγμή που ακούστηκαν τα νέα. Ζητήσαμε συνέντευξη με το διευθυντή της Όλαφ, ήμουν και εκεί παρόν και πρέπει να πω ότι δεν διευκρινίστηκε η κατάσταση, δεν ξεκάθαρη για μένα, πολύ ξεκάθαρη. Το βασικό θέμα ότι είναι ότι δεν είναι δημόσια, δεν μπορεί να δημοσιευτεί η έκθεση της Όλαφ ούτε ε, με τη μορφή εμπιστευτικού εγγράφου. Η Εποπτική Επιτροπή έχει δικαίωμα να δει το κείμενο, την έκθεση και μπορεί να κοινοποιήσει λίγο πολύ τα συμπεράσματα σε αυτή την Επιτροπή. Να μας πει τουλάχιστον αν είναι σωστά τα συμπεράσματα ή αν είναι λάθος. Το πρόβλημα είναι ότι αν διαβιβαστεί στις αρχές της Μάλτας, μπορεί να είναι μακροχρόνια η νομική διαδικασία. Αλλά εμεί έχουμε να αντιμετωπίσουμε πολιτικό θέμα. Ε, έδιωξαν από την πόρτα, έδιωξε ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έναν επίτροπο. Και θα πρέπει να κρίνουμε αν αυτό ήταν κάτι λογικό ή όχι. Και δεν μπορούμε να περιμένουμε δύο-τρία χρόνια να λήξει η νομική διαδικασία. Θα πρέπει τις επόμενες ε, εβδομάδες να διορίσουμε νέο επίτροπο από τη Μάλτα. Θέλαμε να ξέρουμε αν υπάρχει κάποια... Σε... Ε, να, λόγος να δούμε κατά πόσο είναι λογική η παρέτηση του κ. Ντάλη ή όχι. Είναι δεν είναι ικανοποιητική κατάσταση για μας. Έχουμε μόνο αυτά που μας είπε ο Διευθυντής ε, της Όλαφ. Δεν έχουμε κάποια ανακοίνωση της Εποπτικής Επιτροπής. Και πρέπει να περιμένουμε επί μακρόν μέχρι ότου ολοκληρωθούν και αποπερατωθούν οι νομικές διαδικασίες. Θα ήταν πάρα πολύ καλό για μας αν μπορούσαμε να ξέρουμε κάτι παραπάνω από πλευράς ε, Όλαφ, όσον αφορά την έκθεση της Όλαφ. Ευχαριστώ. Ε, πείτε μας εσείς. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Δύο ερωτήματα τέθησαν. Πρώτο, τέθη το πρόβλημα της απουσίας του Γενικού Διευθυντού και ότι δεν μπόρεσε να υπάρξει αντιπαράθεση με αυτά που είπαμε εμείς. Δεν είναι η πρώτη φορά, σας διαβεβαιώ. Δεν είναι η πρώτη φορά που το συζητούμε αυτό. Το συζητήσαμε μακροσκελέστατα με αυτόν. Του στείλαμε επιστολές. Ε, επιμέναμε για καλύτερη συνεργασία διαπραγματευτήκαμε συμφωνήσαμε επί των μεθόδων εργασίας αλλά τα πράγματα δεν είναι τόσο καλά όσον αφορά τον τρόπο λειτουργίας μας και η στελέχωση όπως προαναφέρθηκε πόρο απέχει από το να είναι επαρκής πρέπει να θυμόσαστε ότι εμείς οι πέντε δεν είμαστε μέλη πλήρους απασχόλησης χρειαζόμαστε τη στήριξη προσωπικού που να είναι επαρκές, όχι μόνο από πλευράς ικανοτήτων που είναι, αλλά και σε αριθμό. Και αυτό είναι ένα από τα θέματα που θέταμε. Όσον αφορά την υπόθεση Ντάλι, το δεύτερο θέμα, ο κ. Κέσλερ σας ενημέρωσε και δεν θα μιλήσω, η δική του απόφαση σας ενημερώσει. Σας ενημέρωσε όταν ολοκληρώθηκε η έρευνά του και όταν αποφάσισε να τη διαβιβάσει στις εθνικές αρχές. Όπως είπα, εμείς, και αυτή είναι η δική μας διαδικασία, εμείς είμαστε στην εξή θέση. Η συγγήτρια ακόμα εξετάζει την υπόθεση και πρέπει πρώτα να υποβάλει αναφορά και έκθεση στην Ολομέλεια τη δική μας, που προβλέπεται να λάβει χώρα 22 Νοεμβρίου, τούτου λεχθέντος. Και είναι πολύ σημαντικό να το γνωρίζει κανείς και ίσως να υπάρχουν και κάποιες παρεξηγήσεις από αυτού. Εμείς, η Εποπτική Επιτροπή, δεν είμαστε δικαστήριο. Δεν έχουμε εξουσίες να κρίνουμε κατά πόσο το περιεχόμενο του φακέλου της υποθέσεως που προετοιμάστηκε από την Όλαφ είναι σωστό ή όχι. Είμαστε εκεί και έχουμε σαν αποστολή να παρακολουθούμε το ερευνητικό έργο και αυτό σύμφωνα με τις τη προδιαγραφή και πλήρη σεβασμό ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών. Και ακόμα το τελευταίο τμήμα δεν συμφωνεί με αυτά που θεωρεί ο κ. Κέστερ ότι είναι τα σωστά που πρέπει να γίνονται για μια συνεργασία. Ευχαριστώ. Ο κ. Σέρενχάουζερ είναι επόμενο στο κατάλογο. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ δεν θα επαναλάβω τα ίδια. Συμφωνώ με την κυρία Γκρέσλερ, κατανοώ και τον κύριο Γκάιερ. Όμως η υπόθεση Ντάλι προφανώς επηρεάζει το, την ελεγκτική λειτουργία και το πώς ασκούνται οι αρμοδιότητες ελέγχου. Γιατί θα πρέπει να δούμε την συνεργασία μεταξύ Επιτροπής και Γενικού Διευθυντή της Όλαφ. Είναι δηλαδή μια συγκρουσιακή συνεργασία ή γνήσια συνεργασία. Μήπως κρύβονται και τα δύο μέρη πίσω από ε, παραγράφους και προθεσμίες υπάρχει καλή και λογική συνεργασία. Και γι' αυτό ρωτάω πώς διαμορφώνεται η συνεργασία μεταξύ των, του, του οργάνου ελέγχου και του ίδιου του διευθυντή. Υπάρχουν βαρύνουσες ε, επιπτώσεις ε, μετά από την υπόθεση αυτή ή προϋπήρχαν τα προβλήματα. Επίσης, μιλήσατε για το πρόβλημα του προσωπικού. Δεν αναφέρατε συγκεκριμένα νούμερα. Μπορείτε να μας δώσετε νούμερα. Ε, θα, και ποιος είναι ο σωστός αριθμός για να γίνεται και σωστά η άσκηση των ε, αρμοδιοτήτων σας. Ποιος θα απαντήσει, ο κύριος Ντένολφ. Ναι, μπορώ να απαντήσω. Ευχαριστώ πολύ. Παίρνετε το λόγο μετά εσείς. Λοιπόν, αυτό που θα ήθελα να πω, ευχαριστώντας σας για την ερώτηση, η συνεργασία με την Όλα θα μπορούσε να είναι καλύτερη. Και όσον αφορά την υπόθεση Ντάλι, αν μιλήσουμε για μεθόδου εργασία και πώ πρέπει να εργαζόμαστε, η υπόθεση Ντάλι είναι ακριβώ είναι μία υπόθεση, μόνο μία υπόθεση. Που δέχεται μεγαλύτερη προσοχή από τον τύπο όλα. Συζητούσαμε άλλε υποθέσει. Στην εισαγωγή μου, ελπίζω να θυμόσαστε ότι είπα ότι καταρχά με την κυρία Κρέστη συναντηθήκαμε τον Απρίλιο. Διοριστήκαμε αρχέ αυτού του έτου Ακόμα και τον Απρίλιο είχαμε προβλήματα, πριν ξεσπάσει η υπόθεση Ντάλι. Η υπόθεση Ντάλι σχετίζεται βέβαια με τη συνεργασία, αλλά δεν έχει καμία σχέση ε, σαν γενεσιουργό αιτία. Είναι μία υπόθεση, όπω είχαμε άλλε υποθέσει, όπου εκεί θεωρούμε ότι δεν έχουμε επαρκή συνεργασία. Όσον αφορά τη στελέχωση, το προσωπικό, με τα χαρά σα απαντήσω. Κοιτάξτε, εμεί η Εποπτική Επιτροπή θα θέλαμε να έχουμε λόγο όσον αφορά την πρόσληψη του προσωπικού. Θα θέλαμε να ξέρουμε ποιος εργάζεται για μας. Και προβλεπόταν ότι οκτώ άτομα πλήρους απασχόλησης θα εργαζόταν στο προσωπικό της Όλαφ και τις αρχές του έτους χωρίς να μας συμβουλευτούν, χωρίς να μας ενημερώσουν, ο Γενικός Διευθυντής αποφάσισε να μειώσει τον αριθμό από 8 σε έξι ε, ανθρώπους και όχι με ισοδυναμία πλήρου απασχόληση Τούτου λεχθέντο, έξι άτομα για όλη τη δουλειά που έχουμε που όρο απέχει από το να είναι ο σωστό αριθμό. Γι' αυτό επιμένουμε να έχουμε ξεχωριστό κονδύλι του προπολογισμού για να μπορούμε στο μέλλον να αποφασίζουμε για τη δική μα τελέχωση, να έχουμε ικανού ανθρώπου και να μπορούμε να του προσλαμβάνουμε με τον τρόπο που θεωρούμε σωστό. Διοριζόμαστε από τα τι θεσμικά όργανα. Αν υπάρχει ένα κενό, θα πρέπει να είναι ανοιχτή θέση για όλα τα θεσμικά όργανα. Έτσι ήταν στο παρελθόν. Θέλετε να συμπληρώσετε, κύριε Μπέος, παρακαλώ. Μας πήραν ένα τέταρτο του προσωπικού μας, χωρίς να φταίμε εμείς, γιατί στους κανόνες λειτουργίας μας λέγεται ότι μόνο μετά από γνωμοδότηση δική μας ε, καθορίζεται το προσωπικό. Αλλά δεν υπάρχει τέτοια συμμετοχή μας. Ξέρουμε πώς μπορεί να αποφύγει κανείς έναν έλεγχο αν δεν υπάρχει προσωπικό και χρήματα για αυτόν τον έλεγχο. Ευχαριστούμε λοιπόν πολύ το Κοινοβούλιο που πήρε αυτή την πρωτοβουλία και έγραψε αυτά τα 8 ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης. Να δούμε λοιπόν τι μπορούμε να κάνουμε με αυτή τη δική μας γραμμή του προπολογισμού που εγκρίνεται στην πρώτη ε, ανάγνωση. Να δούμε πώς θα γίνει. Να δούμε μήπως ε, δεν εφαρμοστεί αυτό που ζητάμε. Τώρα κάτι για τον ρόλο της Επιτροπής Εποπτείας αυτής στην αρχή όταν είχαμε αυτή τη συζήτηση για το πώς από μια εξαρτημένη ούκλαφ θα περάσουμε σε μια ανεξάρτητη όλαφ το 1990 είχαμε διαπιστώσει ότι εδώ ακριβώς η Κομισιόν έλεγε θέλουμε ανεξάρτητη Όλα, αλλά που αρχίζει και που τελειώνει η ανεξαρτησία τη, θα το πούμε εμεί το Κοινοβούλιο. Εμεί η Επιτροπή, συγγνώμη. Το Κοινοβούλιο είπε όχι. Όχι, αυτό θα το κάνει ο ανεξάρτητο Γενικό Διευθυντή που θα εκλεγεί και από τα τρία θεσμικά όργανα. Αυτή ήταν η ουσιώδη διαφορά. Οπότε, τι σημαίνει αυτό για την περίπτωση, για μια περίπτωση όπως ε, η περίπτωση Νταλή, που είναι ακριβώς μέλος της Επιτροπής. Οπότε το θέμα της ανεξαρτησίας είναι σαν συναγερμός που αναβοσβήνει. Πόσο ανεξάρτητη είναι η Όλαφ. Είναι όντως ανεξάρτητη. Πόσος χρόνος πέρασε από την καταγγελία μέχρι την αρχή της εξέτασης. Πόσο θα πρέπει να κρατάει συνήθως αυτή η διαδικασία και πώς θα καταλήξει η διαδικασία. Θα υπάρχουν συμπεράσματα, θα εφαρμοστούν Κοιτάξτε, δεν είμαστε δικαστήριο. Αλλά αυτά τα θέματα μπορούμε να τα διαπιστώσουμε, μπορούμε να τα διατυπώσουμε, ούτως ώστε να διαπιστώσουμε εάν όντως λειτουργεί ανεξάρτητα η Όλαφ είτε όχι. Διότι Βεβαίω η, ανεξαρτησία του υπαλλήλου δεν είναι έναντι τη καπνοβιομηχανία. Έναντι τη καπνοβιομηχανία καπνοβιομηχανίας είναι ανεξάρτητος ένα υπάλληλο. Η ανεξαρτησία είναι έναντι τη δική του υπηρεσία. Γι' αυτό χρειάζεται μια ισχυρή εποπτική αρχή. Εάν όμω η εποπτική αρχή δεν είναι καν σίγουρη αν θα τη στείλει ο Γενικό Διευθυντή μια έκθεση για το θέμα αυτό, τότε για ποια ανεξαρτησία μιλάμε. Να δια διευκρινίσω ότι η Όλαφ υπάρχει κίνδυνος να επανέλθει στην αγκαλιά της Κομισιόν από όπου ξεκίνησε. Να της αφαιρεθεί δηλαδή ανεξαρτησία. Είτε θα τηρήσουμε αυτές ε, τις διαδικασίες ελέγχων και ισορροπιών, αλλά πρέπει να συμβάλλουν σε αυτή την προσπάθεια και τα τρία θεσμικά όργανα γιατί ανήκουν και στα τρία και όχι μόνο σε ένα θεσμικό όργανο ανήκουν οι υπηρεσίες της Όλαφ. Χρειαζόμαστε δίκαιο. Χρειαζόμαστε να έχουμε δικαίωμα να παρέμβουμε και όχι παράκληση. Κοιτάξτε, εδώ έχετε μία ανακοίνωση. Η ανακοίνωση όμως αυτή ότι θα γίνει μία έρευνα είναι περισσότερο μαύρη παρά άσπρη. Είναι σαν να είναι παραμύθια. Πρέπει να είναι σαφές. Εάν θέλουμε αποτελέσματα από την εποπτική αρχή πρέπει να εξασφαλίσουμε πλήρη πρόσβαση για μας. Πλήρη πρόσβαση και χωρίς συνθήκες. Δεν μπορεί να ε, ε, εποπτεύσει κανείς κάποιον που δεν του δίνει πλήρη πρόσβαση. Αυτό παρακαλώ να προσέξετε και κατά την τροποποίηση του κανονισμού για την Όλαφ. Να μην υπάρχουν σκοτεινά σημεία. Για παράδειγμα, και εδώ μας διδάσκει κάτι περί περίπτωση Νταλή. Να μην είναι δυνατόν στο μέλλον η εποπτική αρχή να μπορεί να δει ορισμένα έγγραφα μόνο όταν σταλούν και στις εθνικές αρχές. Βεβαίως. Τότε θα περιμένουμε μέχρι που να πεθάνουμε όλοι. Πρέπει να υπάρχουν σαφείς κανόνες. Εσείς μπορείτε να μας ζητήσετε μία ε, έκθεση, ανα πάσα στιγμή. Και για αυτή την περίπτωση. Να είναι όμως κάτι σαφές. Εάν όμως δεν υιοθετούνται και δεν εφαρμόζονται κάποιες διαδικασίες, δεν είναι σαφές ποιος είναι θύμα και ποιος είναι θήτης. Και θύματα... Α, ε, ε, εάν δούμε τι λέει η απόφαση του δικαστηρίου στην περίπτωση Φράνσο Εμπίκ, θα διαπιστώσουμε ότι το θύμα είναι πάντα φορολογούμενος και αυτή η περίπτωση μας απασχόλησε ιδιαίτερα. Κατά τα άλλα, επειδή η διαδικασία είναι ακόμη εν εξελίξη, δεν θέλω να πω τίποτα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει και ο κύριο Τόιρα. Με πολύ πάθος αποφανθήκατε για να τα δούμε πάλι έτσι αντικειμενικά. Το ερώτημα είναι γενικά δεν υπάρχει ενημέρωση για υποθέσεις ακόμα και αν το ζητάτε, δεν ξέρω αν είμαι σαφής. Γενικά μπορεί κανείς να πει ότι δεν υπάρχει ενημέρωση ακόμα και όταν τη ζητάτε. Κύριε Ντένολφο, αυτά που είπε ο κύριος Μπες μπορώ να τα ερμηνεύσω με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή είναι σωστό να πω ότι αν η Επιτροπή Εποπτείας, όχι μονομένα μέλη, ως σώμα η Επιτροπή Εποπτείας, όταν ζητεί πλήρη ενημέρωση ε, για τις έρευνες και τα αποτελέσματα των ερευνών του Όλαφ ε, δεν τη λαμβάνει αυτή την ε, πλήρη ενημέρωση. Μπορώ, είναι σωστή η ερμηνεία μου. να, προσθέσω κάτι κύριε Πρόεδρε. Στα αγγλικά θα το πω. Μου είναι ευκολότερο. το πρώτο οκτάμινο μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου, δεν θυμάμαι ακριβώς την ημερομηνία, αλλά περίπου εκείνη την περίοδο, δεν είχαμε επαρκή πρόσβαση στους φακέλους όταν ζητούσαμε και συχνά όταν ε, είχαμε την πρόσβαση ήταν υπερβολικά αργά. Η κατάσταση ήταν εντελώς μη ικανοποιητική. Ε, κάναμε διαμακρών συζητήσεις με τον Γενικό Διευθυντή για να εκφράσουμε τη δυσαρέσκειά μας και του στείλαμε δυο φορές επιστολή όπου λέγαμε ότι αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση δεν μπορούμε να αναλάβουμε καμία ευθύνη για αυτά που πρέπει να πράξουμε, γιατί δεν μπορούμε να πράξουμε και θα απευθυνθούμε στα θεσμικά όργανα για να εξηγήσουμε την κατάσταση. Από τότε βελτιώθηκαν τα πράγματα. Υπήρξε κάποια βελτίωση, δηλαδή τώρα έχουμε μια διευθέτηση για την εργασία μας, εγγράφος, που όπως είπε και ο Πρόεδρος βασίζεται σε μια πρόταση που ε, έκανε ο Ευρωπαίος Επόπτης ε, Προστασίας Δεδομένων, γιατί η διαφορά μας ουσιαστικά αφορά το εύρος της προστασίας προσωπικών δεδομένων. Είναι νομικό το πρόβλημα. Τώρα βρήκαμε μια μέθοδο εργασίας με τρία βήματα, δεν θα τα εξηγήσω, πάντως το τελευταίο βήμα προβλέπει ότι, ότι αν δεν ικανοποιηθούμε από τις πληροφορίες που λάβαμε στα δύο προηγούμενα βήματα, θα ζητήσουμε πλήρη πρόσβαση στο φάκελο. Και υπ' αυτή την έννοια υπάρχει ακόμα μια διαφορά μεταξύ μας και με το Γενικό Διευθυντή, γιατί εκείνος λέει ότι πρέπει να ε, μια πλήρη αιτιολόγηση για να έχουμε την πρόσβαση και ότι εκείνος επιφυλάσσεται του δικαιώματος να μην δώσει πρόσβαση. Ο, ήδη αναφέρθηκε ένα παράθεμα από αυτά που είπε ο, Γενικός, από, αυτά που είπε ότι εάν κρίνουμε εμείς ότι πρέπει να έχουμε πλήρη πρόσβαση γιατί αλλιώς δεν μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας, τότε πρέπει να μας χορηγηθεί πλήρης πρόσβασης. Οπότε εδώ υπάρχει ακόμα μια διαφορά απόψεων. Και νομίζω ότι είναι σωστό να πούμε ότι η γενικότερη κατάσταση σε ό,τι αφορά την πρόσβαση είναι τώρα γενικά πιο ικανοποιητική από ό,τι ήταν στο παρελθόν. Γιατί πολλές φορές μας έλεγαν ένα σκέτο όχι. Εις ό,τι αφορά το όμως την ικανοποιητική εφαρμογή αυτής της ε, λύσης που βρέθηκε, αυτής της διευθέτησης, ακόμα πρέπει να γίνει δουλειά. Δεν είναι όμως ε, σωστό να πούμε, δεν θα είμαστε δίκαιοι αν λέγαμε ότι η κατάσταση είναι τόσο άσχημη όσο ήταν το προηγούμενο οκτάμινο. Ο κύριος Εντερόλφ. Μπορώ να προσθέσω κάτι σε αυτά. Πράγματι, Τώρα εργαζόμαστε βάσει αυτή τη ρυθμίσεω. και είμαστε στα πρώτα δύο βήματα. Πρώτο βήμα, δειγματοληψία παραδείγματο Όσον αφορά το πρώτο βήμα, είναι σημαντικό αυτό που σας είπε ο Χέρμπερτ. Το μαύρισμα κάποιων τμήματων των εγγράφων είναι τόσο εντυπωσιακό που δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα με το έγγραφο. Το συζήτησα με το Γενικό Διευθυντή χθες και μου είπε τα ονόματα και οι εταιρείε πρέπει να μαυριστούν, να καλυφθούν. Τα υπόλοιπα όχι όμως. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έχει καλυφθεί για την ώρα. Αν πάμε πάλι στην ομοδότηση του EDPS, την ίδια σελίδα, σύμφωνα το άρθρο 2,3, Όσον αφορά όταν αποδεικνύεται ότι είναι ανεπαρκή τα στοιχεία και εμποδίζουν την εποπτεία και η εναρμόνιση του φακέλου από πλευρά όλαυση απαιτεί δυσανάλογη προσπάθεια, μπορεί να έχει ε, πλήρη πρόσβαση η υποπτική αρχή. Εάν υπάρχουν μεγάλοι φάκελοι, δεν χρειάζεται να καλυφθούν κάποια στοιχεία, πρέπει να μας εμπιστευτούν. Αυτή τη συζήτηση έχουμε τώρα. Ε, δεν προχωρούν ομαλά τα πράγματα, είναι δύσκολα, θα μπορούσαν να είναι καλύτερα και δεν είμαστε σε θέση να κάνουμε τη δουλειά μας σωστά όπως έχουν τα πράγματα. ως μας, ε, έχει, μας έχουν διορίσει, μας έχουν καθορίσει το πλαίσιο των εργασιών μας τα θεσμικά όργανα. Ευχαριστώ κύριε Τίμπερμαντς, ε, ε, μας δώσατε πολύ σημαντικές πληροφορίες. Ε, συνοψίζοντας, από ό,τι κατανοούμε, έχετε την εντύπωση ότι παίρνετε πολύ καθυστερημένα τους φακέλους, σας δίνουν πολύ λίγες πληροφορίες Λίγες πληροφορίες, καθυστερημένα, πολύ καθυστερημένα και αυτό πρέπει να ερευνήσουμε είναι το θέμα της προστασίας των δεδομένων. Διότι από ό,τι κατάλαβα μέχρι τώρα, η Επιτροπή Εποπτείας είναι ένα απόσπαστο τμήμα του καθεστώτος της Όλαφ. Εάν η Όλαφ μπορεί να πάρει τα στοιχεία, τότε και η Επιτροπή Εποπτείας πρέπει να έχει τα στοιχεία, διότι υποχρεούστε ε, να διατηρήσετε τα στοιχεία εμπιστευτικά. Ίσως είναι νομικό πρόβλημα προς διερεύνηση. Πρέπει να το διερευνήσουμε περαιτέρω. Κύριε Τίμπερμαντς, είπατε ότι αυτό δεν είναι σωστό. Κάτι είπατε πάνω. Είχα μακρά συζήτηση με τον ε, επόπτη προστασία των δεδομένων πριν από μερικές εβδομάδες για αυτό το θέμα και μου εξήγησε κάποια πράγματα. Και το έλεγξα αυτό και στα κείμενα. Και είναι σωστό αυτό που μου είπε. Μου είπε ότι και εντό ενός θεσμικού οργάνου, ενός φορέα, η μεταβίβαση πληροφοριών, στοιχείων, εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογή των κανόνων του κανονισμού, των άρθρων του κανονισμού. Είναι η χορήγηση πληροφοριών κατά ανάγκη ενημέρωση. Need to know. Αν δείτε στην ε, Γενική Διεύθυνση Κόμπ, βλέπετε ότι όλοι όσον αφορά όλα τα μέλη της Γενικής Διευθύνσεως περί ανταγωνισμού, έχει πρόσβαση στους φακέλους περί Μόνο αυτοί που έχουν λόγους να έχουν πρόσβαση, δέχονται την πρόσβαση. Αυτό είναι κάτι που προστατεύεται σύμφωνα με τους κανόνες της προστασία των δεδομένων. Ακόμα και εντός της Επιτροπής Εποπτείας, που είναι εντός της Όλαφ, είτε είμαστε εσωτερικό ή εξωτερικό φορέα, αν είμαστε εσωτερικό ή εξωτερικό φορέα τη Όλαφ, και αυτό το συζητήσαμε, δεν σα κουράσω με αυτό, αλλά και μεταφορά πληροφοριών, μεταβίβαση πληροφοριών εντός της Όλαφ προ εμά είναι κάτι που προστατεύεται εάν πρόκειται περί προσωπικών δεδομένων. Αυτό ήθελα να πω. Ευχαριστώ για τη διευκρίνηση. Δεν αμφισβητεί κανείς την αρχή αυτή, νομίζω. Ε, όχι, όχι η κυρία Γκρέσλε. Όχι, για το θέμα προστασίας δεδομένων θέλω να πω κάτι. Η προστασία δεδομένων δεν ε, προέρχεται από τη γραμματεία της ε, Κομισιόν. Πώς γίνεται συστηματικά να διαβιβάζονται οι κλεισμένες ε, έρευνες σε αυτό το σώμα. Εμείς είχαμε μιλήσει για παραβίαση. Πιστεύω ότι έχουμε να κάνουμε με μία ε, ε, διαδικασία που αποφασίζει ο Γενικός Διευθυντής πότε είναι καλή η προστασία δεδομένων και πότε πρέπει να την προστατεύουν. Εκείνοι που δεν χρειάζονται την πληροφορία, η Γενική Γραμματεία, μπορούν να τη λαμβάνουν. Εκείνοι που τη χρειάζονται, όχι. Αυτή η αυταρέσκεια δεν με βρίσκει σύμφωνη, δεν την ε, παραδέχομαι. Βεβαίω είναι θέμα πάντοτε η προστασία δεδομένων. Αλλά το κομικό είναι ότι δεν είναι το ίδιο προβληματικό για όλου και το ίδιο ε, αφορά αυτές τις κλεισμένες ε, ε, έρευνες και τις σχετικές εκθέσεις. Εγώ δεν είμαι διατεθειμένη να ακούσω επιχειρήματα τα οποία θα φρενάρουν τη σωστή διαδικασία, ιδιαίτερα όταν είναι τόσο ισχνά και δεν αναφέρομαι σε εσά προσωπικά, όταν είναι τόσο ισχνά όπως αυτά που αναφέρονται. Ευχαριστώ πολύ. Άφησα να μιλήσει η κυρία Γκρέσλε γιατί είναι η συγγήτρια. Κυρία Πινιό και μετά η κυρία Αντρέασεν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν θα εκφραστώ επί της συγκεκριμένης ε, περιπτώσεως, αλλά ε, σε σχέση με αυτά που ήδη υπόθηκαν. Θεωρούμε ότι το θεμελιώδες θέμα είναι να καθορίσουμε τι πληροφόρηση χρειαζόμαστε για να μπορούμε και με πλήρη και με αυστηρό τρόπο να είμαστε σε θέση να επιτελέσουμε την αποστολή μας, να ελέγξουμε και να αποτιμήσουμε σε τι βαθμό η Όλαφ παίζει το ρόλο της και όσον αφορά την αμεροληψία και όσον αφορά την αποτελεσματικότητα και φυσικά όσον αφορά το σεβασμό κατά, τον, ε, κατά τη διεξαγωγή των ερευνών της, ε, των σωστών διαδικασιών και διοικητικών εγγυήσεων. Είναι σαφές ότι αυτή η αρμοδιότητα ελέγχου σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε πρόσβαση στην πληροφόρηση στο βαθμό που θεωρούμε ότι έχουμε ανάγκη από πληροφόρηση για να μπορούμε να παίξουμε αποτελεσματικό το ρόλο μας. Είμαστε υπεύθυνοι για τη δουλειά μας, όχι έναντι του Γενικού Διευθυντή της Όλαφ, αλλά έναντι των θεσμικών οργάνων που μας διόρισαν. Πιστεύουμε λοιπόν ότι δεν θα ήταν δυνατόν ο οργανισμός που ελέγχουμε να υπαγορεύει σε τι βαθμό θα μας ενημερώσει για να κάνουμε τη δουλειά μας. Το θεμελιώδες θέμα που θα θέλαμε να διατυπώσουμε σήμερα ήταν αυτό ακριβώς ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Πινιόν. Επόμενη η κυρία Ανδρέασεν. Ευχαριστώ. Κύριε Ντένολφ, είπατε ότι ο κύριος Κέσλερ δεν σέφεται τους ε, κανόνες του. Αλλά και τους δικούς σας. Πώς εκπονήθηκαν αυτοί οι κανόνες. Θα ήθελα να μάθω εάν κάποιοι από αυτούς τους κανόνες συγκρούονται με τον κανονισμό της ίδιας της Όλαφ. Εμείς συμμετείχαμε στην ε, εκπόνηση του κανονισμού του Όλαφ αλλά δεν συμμετείχαμε στην ε, διατύπωση των κανονισμών για τη δική σας εσωτερική λειτουργία. Θέλω να μου πείτε πώς εκπονήθηκαν οι κανόνες λειτουργίας σας και αν υπάρχει ενδεχόμενο σύγκρουση συμφερόντων. Πώς μπορεί ο κύριος Κέσλερ να μην σας επιτρέπει να έχετε περισσότερο προσωπικό. Δεν ξέρω αν κατάλαβα καλά. Μας είπατε ότι εκείνο δεν έχει επαρκές προσωπικό για να κάνει τι έρευνε του ή εσείς ως εποπτική αρχή δεν έχετε επαρκέ προσωπικό για τις δικές σας έρευνες. Γιατί αν είστε εσείς που δεν έχετε επαρκές προσωπικό, δεν νομίζω ότι ο Γενικός Διευθυντή τη Όλαφ είναι αρμόδιος για να εγκρίνει το προσωπικό σας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει το προσωπικό σας. Εκείνη έχει τον προπολογισμό. Δεν ξέρω τι ακριβώ συζητάμε. Θέλω κάποιε διευκρινήσει. Με ποιο τρόπο μπορεί να σα πει ότι δεν μπορείτε να προσλάβετε επιπλέον προσωπικό. Νομίζω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρεμβαίνει εδώ. Τώρα, για την περίπτωση Ντάλι. Ο μόνος ρόλος που έχουμε εμείς εδώ είναι να διασφαλίσουμε ότι ο ΛΑΦ ακολούθησε την ορθή διαδικασία. Δεν θα επισέλθουμε στις δικές σας συγκρούσεις με την Όλαφ. Εμείς πρέπει να ελέγξουμε εάν η Όλαφ ακολούθησε την σωστή διαδικασία. Δεν θα κρίνουμε τον Τάλι. Αν θέλετε να μάθετε για την ε, παρέτησή του και την ε, αναστολή ε, άσκηση των καθηκόντων του, την διαθεσιμότητά του, αυτό είναι θέμα του Πειθαρχικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν θα συζητήσουμε εμείς με την Όλαφ για πειθαρχικά θέματα. Όσον αφορά την ανεξαρτησία της Όλαφ. Εδώ και πολύ καιρό έχω καταλάβει ότι ποτέ η Όλαφ δεν θα είναι εντελώς ανεξάρτητη εφόσον ε, τις εκθέσεις της τις κάνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νομίζω ο κύριος Μπέος ξέρει για τα σχόλια που έχω κάνει εδώ για και 10 χρόνια για αυτό το θέμα. Ευχαριστώ κύριε Αντριάνσεν, λέει ο πρόεδρος. Ο κύριος Ντένοφ. Ναι, τέσσερα θέματα. Ανεξαρτησία της Όλαφ. Κοιτάξτε, η ανεξαρτησία της Όλαφ ε, Είναι δυσχερές καθήκον, αλλά πρέπει να το ελέγχει κανείς, να το εποπτεύει κανείς για το προσωπικό. Το διοικητικό προσωπικό της Όλαφ. Επιτηρούνται από την ε, Επιτροπή. Οι ερευνητικές λειτουργίες της Όλαφ ερευνάται μόνο από μας. Να το διευκρινίσουμε αυτό. Θα πρέπει λοιπόν να μπορούμε να κάνουμε σωστά αυτή τη δουλειά. Και μας διορίζουν όλους και τα τρία θεσμικά όργανα, γιατί είμαστε ειδήμονε στον τομέα μας. Δηλαδή, είμαστε αρκετά ειδήμονε για να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας, εάν μας δώσουν τα επαρκή μέσα. Ευχαριστώ για την παρατήρηση. Ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις σα για την υπόθεση Ντάλι. Τώρα για τον αριθμό συνεργατών, υπαλλήλων. Η Όλαφ μα δίνει το προσωπικό τη. το προσωπικό μα. Οπότε εμεί ως Επιτροπή Εποπτείας μπορεί να φαίνεται αστείο για τους Βατανούς μπορεί να νομίζετε ότι είναι κρίκετ. Όταν είστε μέσα είστε έξω και όταν είστε έξω είστε μέσα. Αυτή είναι η έκφραση από το κρίκετ. Είμαστε εκτός Όλαφ όταν τη βολεύει και εντός Όλαφ επίσης όταν τη βολεύει. Είναι θέμα οπτικής γωνίας. Πρέπει να διευκρινιστεί. Να διευκρινιστεί διότι δεν πρόκειται περί αθλοπαιδιών. Τώρα το επίπεδο του προσωπικού. Το προσωπικό μας είναι τμήμα της Όλαφ. Η Όλαφ έχει περίπου 500 άτομα. Εμείς έχουμε 8. 8 για να επιτηρήσουμε την Όλαφ. Τώρα έχουμε μείνει στους 6. Αλλά όχι 6 πλήρους απασχόλησης. Θα έπρεπε να έχουμε 6 ισοδύναμα, ενώ έπρεπε να έχουμε 8 ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης. Δηλαδή να έχουμε τον προϋπολογισμό για 8 θέσεις πλήρους απασχόλησης. Γι' αυτό θέλουμε την υποστήριξή σας. Δώστε μας τη δική μας γραμμή του προπολογισμού και με τις πιστώσεις αυτές θα μπορούμε να έχουμε 8 ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης. Βεβαίως, ο Γενικός Διευθυντής Κέσλερ αποφασίζει για το προσωπικό μας. Μπορεί να αποφασίσει πόσους θα έχουμε. Να αφαιρέσει κάποιον όταν τον βολεύει και να τον αντικαταστήσει με κάποιον άλλον. Όπως και κάνει. Μπορούμε να αμφισβητήσουμε την απόφαση, αλλά σε τελευταία ανάλυση αυτός αποφασίζει. Ούτως έχουν τα πράγματα. Και πρώτο και ίσως το πιο σημαντικό για τους ε, κανόνες λειτουργίας μας, τον εσωτερικό κανονισμό μας. Επιβεβαιώθηκαν από την προηγούμενη Επιτροπή το 2011, από τη δική σας Επιτροπή. Και θέλω να πω ότι με εντυπωσιάζει ιδιαίτερα αυτό. Κατά τη γνώμη μου, οι κανόνες αυτοί είναι πολύ καλοί. Πολύ ορθά διατυπωμένοι. Με βάση τον κανονισμό διατυπώθηκαν γι' αυτό. Και ό,τι περιέχουν βασίζεται στον κανονισμό 1073. Τι έκανε η προηγούμενη Επιτροπή Εποπτείας. Έστειλαν αυτόν τον ιστορικό κανονισμό στα τρία θεσμικά όργανα. Και τους μελέτησαν τα τρία θεσμικά όργανα και δεν έκαναν παρατηρήσεις. Και επιπλέον δημοσιεύθηκε στην επίσημη εφημερίδα της Ένωσης. Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι ότι ο Γενικός Διευθυντής που ήδη είχε αναλάβει τότε δεν συμφωνούσε με αυτούς τους κανόνες. Εάν δεν συμφωνούσε, γιατί δεν αντέδρασε τότε. Ευχαριστώ πολύ. Τελευταίος, ε, αν, τελευταία, εάν δεν παρέμβλεψα κανέναν, η κυρία Γκρέσλε. Επανέρχομαι σε δύο-τρία θέματα, συγγνώμη. Καταρχήν, Γιένς, το θέμα της αντιμετώπισης της Επιτροπής Εποπτείας και των δυνατοτήτων εργασίας του για μένα είναι το πιο σημαντικό θέμα. Αυτή είναι η ουσία της σημερινής μας συνάντησης. Το ωραίο στην υπόθεση Ντάλι όμως είναι ότι είναι από τις λίγες υποθέσεις που μας ε, γνωστοποιήθηκαν. Οπότε ε, υπάρχει ένα μεγάλο ε, έλλειμμα ενημέρωσης και το ενδιαφέρον είναι ότι ξαφνικά έχουμε ερωτήσεις που αφορούν την ίδια τη διαδικασία στην Όλαφ. Δηλαδή, ποιο είναι το ερώτημα. Πρόκειται για μια ενορχιστρωμένη ε, επίθεση κατά, που σπηλώνει κάποιον και που καλύπτεται ή δεν αποκαλύπτεται ε, ε, όπως πρέπει από την Όλαφ. Ή, δηλαδή, έχουμε μόνο καπνό ή όπου είναι καπνός είναι και φωτιά. Αυτά μας κάνουν να, μπορούμε. να Και είναι πολύ σημαντικό γιατί αυτό αφορά τη λειτουργικότητα της ίδιας της Όλαφ. Βέβαια, ε, βλέπω ότι και η ομάδα σου το βλέπει το ίδιο. 20 λεπτά μετά την συνάντηση που είχαμε στην Κοκομπή, ο πρόεδρος της Επιτροπής σου έκανε ανακοίνωση στον τύπο, δήλωση στον τύπο, που λέει ότι τώρα φαίνεται ότι η κατάσταση δεν αντιμετωπίστησε σωστά από τον πρόεδρο της Κομισιόν και τον Γενικό Διευθυντή της Όλοφ. Και μετά λέει μήπως επρόκειτο για κάποια ε, ε, συνωμοσία. Ε, ο δικός μου πρόεδρος δεν θα, της ομάδας μου δηλαδή χωρίς να με συμβουλευτεί δεν θα είχε προβεί σε τέτοια δήλωση πάντως αυτό πρέπει να το πω όχι γιατί χρειάζεται πραγματικά να έχουν και οι, τα ε, μέλη ε, κάποια ισχύ τώρα πρέπει να δούμε την έκθεση του, της Όλαφ και να δούμε και το συνοδευτικό του Γενικού Διευθυντή προς τον ε, Πρόεδρο της Κομισιόν, του Γενικού Διευθυντή προς τον Πρόεδρο. Αυτά πρέπει, σε αυτά πρέπει να επιμείνουμε κύριε Πρόεδρε, γιατί αλλιώς δεν θα προχωρήσουμε σε αυτή την υπόθεση και δεν θα ξέρουμε γιατί πρέπει να κάνουμε. Να μας πείτε και για την επόμενη συνεδρίαση πότε θα ε, την κάνουμε για να ενημερωθούμε από εσάς. Τι αποτελέσματα είχαν οι έρευνές σας. Ε, η έκθεση Όλαφ που δεν, έχει, ε, δεν είναι νομική ε, πριν από τη Μάλτα, εάν συμφωνεί η Μάλτα μπορούμε να την έχουμε. Αυτό δεν νομίζω ότι είναι ε, σημαντικό γιατί αλλιώς θα έπρεπε να παρακαλούμε την κάθε ερευνητική επιτροπή, επιτροπή έρευνας. Εγώ πάντως, α, θα ήθελα και μια εναλλακτική. Ε, θα μπορούσα να, προβλέψω και εναλλακτική μέθοδο. Ε, πάντως μου αφήνει μια άσχημη γεύση όλη αυτή η υπόθεση. Ε, έχουμε εδώ έναν ε, αυταρχικό γενικό διευθυντή, ο οποίος δεν μπορεί να αφήσει το σώμα που συγκροτήσαμε να εργαστεί και φαίνεται ότι δεν είναι δυνατόν να πιστή. Εγώ παρακάλεσα και τον ε, ε, κύριο Σίμετας και μου υποσχέθηκε ε, ότι θα μιλήσει και μου είπε ότι μίλησε με τον αρμόδιο, αλλά η κατάσταση αυτή δεν πρέπει να συνεχιστεί. Για το προσωπικό θα πρέπει να γίνει διαγωνισμός και θα πρέπει εσείς να είστε υπεύθυνοι, να έχετε βαρύνοντα λόγο στην επιλογή του προσωπικού. Δεν μπορεί δηλαδή να αποδέχεστε όποιον σας βάλουν εκεί. Ε, υπάρχει θέμα εμπιστοσύνη, υπάρχει θέμα ποιότητα τη δουλειά που θα γίνεται και η γραμματεία κάνει πολύ κρίσιμη δουλειά. Είναι μια ε, υπόθεση που θα πρέπει να την ε, πάρουμε στα σοβαρά και να πιέσουμε. Και παλιά έτσι λειτουργούσε και έτσι πρέπει να ξαναλειτουργήσει. Έπειτα, η πρόσβαση από, εσά σας στο σύστημα διαχείρισης των υποθέσεων. Σαφές, χωρίς αυτά, αυτές τις γελίες ε, καλύψεις των μισών κειμένων υπάρχουν περιπτώσεις και υποθέσεις που πρέπει να τις δείτε. Και βλέποντας τα καθήκοντά σας και τα καθήκοντα που θα σας ανατεθούν από τον νέο κανονισμό, πώς θα μπορέσετε να τα ασκήσετε, διαρωτώ με, χωρίς ε, σωστές ρυθμίσεις και κανόνες λογικούς. Επίσης νομίζω ότι ήρθε η ώρα να βελτιωθεί γενικότερα το κλίμα και εμείς στην Επιτροπή μας θα πρέπει να ασχοληθούμε εντατικά με το, την Όλαφ γιατί ορισμένα ε, προβλήματα δημιουργούν αντίκτυπο πολύ αρνητικό. Επίσης κάτι πολύ σημαντικό. Σε αυτή την πολύ δύσκολη υπόθεση Ντάλι όπου βλέπουμε περίεργες εξελίξεις σε πολλά επίπεδα ε, βέβαια και εσείς ε, κύριε Κέμπριτς είστε εδώ ε, ίσως θα έπρεπε να πούμε κάτι και για το δικό σας το ρόλο στην υπόθεση αυτή θα με ενδιέφερε γιατί εσείς ε, είστε υπεύθυνο, είστε ο συνομιλητής από τη Μάλτα της Όλαφ ε, υπάρχει από αρχές Ιουλίου η υπόθεση αυτή νωρίς πρέπει λοιπόν να υπάρχει μια επαφή βλέπουμε ε, υπάρχει πρόβλημα ε, συνεργασίας μεταξύ ελέγχοντος και ελεγχομένου. Αυτό αποδυναμώνει και την Επιτροπή Εποπτείας. Και αυτό δεν είναι καλό, εγώ δεν το θέλω καθόλου. Καλό είναι λοιπόν να μας πείτε και τη γνώμη σας εδώ. Δεν μπορούμε να κρατήσουμε απ' έξω από τις εργασίες της ε, Όλαφ και της ε, Επιτροπής Εποπτείας στην υπόθεση Ντάλι, γιατί είναι η κορυφή του παγόβουνου, αναφύονται πολλά ερωτήματα. Και ε, νομίζω ότι και εμείς αποτελεσματικές πιέσεις θα πρέπει να συνεχίσουμε να ασκούμε και να δούμε και τον Γενικό Διευθυντή και πώς θα μπορέσουμε να τον πείσουμε, να τον πιθαναγκάσουμε σε μια σωστή συνεργασία με όλους τους ε, ε, ενεχομένους. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Εντάξει, αυτή ήταν ε, η καταληκτική τοποθέτηση της εισηγήτριας με κάποιες πολιτικές ε, αξιολογήσει αλλά και κάποιες ερωτήσεις. Δεν ξέρω αν θέλετε ω Εποπτική Επιτροπή να πάρετε το λόγο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την υποστήριξη που μας δίδετε σε αυτό το, στην αντιμετώπιση του προβλήματος. Ζητούσαμε στήριξη σε τέσσερις διαφορετικούς τομείς και τώρα είναι η χρυσή ευκαιρία που έχουμε μπροστά μας, ενώ το νέο κανονισμό. Ήδη δώσατε κάποια άποψη από αυτού συμβουλή, αλλά θα ήμασταν πολύ χαρούμενοι αν γινόταν σεβαστή όλη, όλες οι διατάξεις του εσωτερικού κανονισμού και αν αυτό συμπεριλαμβανόταν ή δυνατόν ο σεβασμός του εσωτερικού κανονισμού. Παρ' όλα αυτά είμαι πολύ ικανοποιημένο διότι μπορώ να στείλω επίσημα στην Κοκοπίου αυτά τα τέσσερα σημεία και να πω ότι θα ζητούσαμε την υποστήριξή σας. Θα ενθαρρύναμε την υποστήριξή σας Στη διακριτική σας ευχέρεια είναι, αν θέλετε βέβαια, να κάνετε κάτι τέτοιο. Όσον αφορά τη θέση ενός μέλους της Επιτροπής Εποπτείας, από αυτά που συζητούσαμε και από αυτά που γνωρίζαμε, που γνωρίζουμε μάλλον, από αυτά που μας είπαν, ενημερωθήκαμε για το ότι ίσως να είμαστε σε κάπως ευαίσθητη θέση. Και ε, ε θα αφήσω την ε, η συνάδελφο να εξηγήσει την ευαισθησία του θέματος αφορά την υπόθεση Ντάλι. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ για αυτά που είπατε. Όπως γνωρίζετε, στις 17 Οκτωβρίου εκλήθη η, Επιτροπή Εποπτείας να ενημερώθηκε για την υπόθεση Νταλή. Την επόμενη, στις 18 του μηνός, έστειλε επιστολή σε όλα τα μέλη και είπα θα αποσυρθώ από την υπόθεση, διότι υπάρχουν αρκετοί ικανοί άνθρωποι στην υπόλοιπη ομάδα μου και μπορούν να ασχοληθούν, να εφαρμόσουν ε, με τις εγγύσεις και να εξετάσουν τι έκανε και τι δεν έκανε η Όλαφ στην υπόθεση Νταλή. Γιατί το έκανα αυτό. Όταν ζήτησα να γίνω μέλος της Επιτροπής Εποπτείας, νομίζω ότι ήταν Δεκέμβριο του 2011, παρουσίασα στα τρία θεσμικά όργανα, όπως και οι συνάδελφοί μου, ένα βιογραφικό σημείωμα. Και σαφώς το βιογραφικό μου λέει ότι είμαι η Γενική Διευθύντρια. Ήμουν τότε έτσι Γενική Διευθύντρια της, του τμήματος της Διευθύνσεως Εσωτερικής Έρευνας και Εποπτείας και που λογοδοτεί στην Εποπτική Επιτροπή ε, και ε, όπου λογοδοτεί και στο Υπουργό στη Και αυτός λογοδοτεί στον ε, Πρωθυπουργό. Και αναφέρεται ότι υπήρχε εμπειρία από το Μάιο του 2008. Ποια ήταν η εμπειρία μου από το 2008 μέχρι σήμερα εξηγούσα ποια ήταν τα καθήκοντά μου για όσον αφορά τους εσωτερικούς ελέγχους και τους οικονομικές έρευνες στην δημόσια δίκηση της Μάλτας αφορούσε, αφορούσε 5,2 δις το 2011. Πέρα αυτό, τις υποχρεώσεις που είχαμε για να συμμορφωθούμε ως ελεγκτικός φορέας και ελεγκτική αρχή όσον αφορά τα προεντεξιακά κονδύλια ταμεία συνοχής, διαθωτικά ταμεία, ε, εδαφική ε, ε, συνεργασία, αλληλεγγύη, διαχείριση μεταναστευτικών ροών και όλα τα προγράμματα και άλλους πόρους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Ελέγχαμε. Και η διεύθυνση της οποίας ήμουν επικεφαλής είναι και ο φορέας διαπίστευσης όσον αφορά το ειδικό τμήμα που ασχολείται με όλα τα γεωργικά κονδύλια, γεωργικούς πόρους. Και αυτά ήταν τα βασικά μου καθήκοντα έναντι των ΑΦΚΟ, αυτά που αποκαλεί όλα ΑΦΚΟ, που είναι μια υπηρεσία συντονισμού κατά πολέμησης των απατών. Όλες οι χώρες ως το 2003 έπρεπε να ε, συνάψουν συμφωνία για διοικητική συνεργασία μεταξύ Όλαφ και Ευρωπαϊκής Επιτροπής και κρατών μελών και υποψηφίων κρατών μελών τότε. Δηλαδή κάθε χώρα θα διόριζε συντονιστική υπηρεσία που θα συντόνιζε και θα βοηθούσε την Όλαφ όταν διενεργούσε επιτόπιους ελέγχους στη χώρα και όταν ζητούσε η χώρα σύμφωνα με τον 1073 του 99 αν το διεξαγωγή έρευνας στη συγκεκριμένη χώρα ή μπορούσε να ζητηθεί να δώσει η χώρα περαιτέρω πληροφορίες. Να σας εξηγήσω λοιπόν τώρα ποιος ήταν ο ρόλος αυτής της μονάδας, της ΑΦΚΟ, που ήταν μια μικρή μονάδα στη διεύθυνση, που ήταν που ενημέρωνε κάθε τριμηνό, παρήχε έναν κατάλογο που αφορούσε τα διαθετικά ταμεία και τις πολιτικές ε, συνοχής. Αυτοί που διαχειριζόταν τους πόρους ενημέρωναν την αρμόδια αρχή ελέγχου για τα σταλίες Μα έστελναν αυτές τις ε, έκθεσει και τροφοδοτούσαμε τις πληροφορίε στο σύστημα ελέγχου για τα σταλίες τη Όλαφ. Αυτό ήταν το βασικό έργο αυτών των υπηρεσιών ελέγχου, των ΑΦΚΟΣ και ήταν παρόμοια προσέγγιση σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πέραν από αυτό, από το 2004 και πέρα, και ήμουν εκεί το 2004, μετά το 2004 λοιπόν, έκανε τέσσερις έρευνες η Όλαφ στη Μάλτα όταν λέω τέσσερις, τι εννοώ. Ζητήθηκε ε, να ε, υπάρξει βοήθεια σε τέσσερις έρευνες. Δηλαδή, μία έρευνα το πολύ κάθε δύο χρόνια. Εδώ συμπεριλαμβάνεται προφανώς και υπόθεση Ντάλι. Όπως είπα τότε, ήμουν επικεφαλής αυτής της μονάδας και έλαβα τηλεφώνημα και μου είπαν ότι καταφθάνει η Όλαφ στη Μάλτα και βέβαιως πρέπει να ενημερώσουν τις επικεφαλής της υπηρεσίας μας δεν δόθηκαν λεπτομέρειες. Ήρθαν λοιπόν στο γραφείο μου 4 Ιουλίου, πράγματι, μας έδειξαν ότι υπήρχαν εικασίες για κακή διαχείριση διαθωτικών ταμείων από κάποιον οικονομικό φορέα της Μάλτας και μας είπαν να διενεργήσουμε επί ότι έπρεπε να διενεργήσουν επιτόπου έρευνες. Εμείς τους δώσαμε, φροντίσαμε για την επιμελητία, τους δώσαμε διευθύνσει κλπ. Και πήγαμε εκεί ως παρατηρητές. Θεωρήσαμε ότι ως χώρα όταν έρχεται η Όλαφ στη Μάλτα πρέπει να παρατηρούμε τα τεκτενόμενα. Μετά από αυτό κάποιος προσεκλήθη για μία συνέντευξη και ως είναι πρακτική σε όλες τις έρευνες της Όλαφ που διενεργούνται στη Μάλτα εξασφαλίσαμε να είναι κάποιο εκεί να παρατηρεί την όλη συνέντευξη. Γιατί? Γιατί αφορούσε Μαλτέζο υπήκο, διενεργόταν αυτή η συνέντευξη στη Μάλτα βάσει του εθνικού δικαίου και θέλαμε να υπάρχουν τα απαραίτητα διαδικαστικά χέγγια. Άλλη μετέτε συνέντευξη έγινε 5 Σεπτεμβρίου, θυμάμαι σωστά, όπου εκεί ξανά μα ζητήθηκε να παριστάμεθα ω παρατηρητέ και η μόνη άλλη εμπλοκή της ε, συντονιστικής υπηρεσίας καταπολέμησης των απατών που είχε υπηρεσία αυτή σε αυτή την έρευνα και καταλαβαίνετε ότι δεν μιλάμε για εθνική έρευνα αλλά για έρευνα Όλαφ. Λοιπόν, η μόνη μας εμπλοκή ποια ήταν. Όσον αφορά τη διοικητική συνεργασία και τις σχετικές διευθετήσεις, εμείς σαν ΑΦΚΟΣ, αν μας ζητηθεί από την Όλαφ να δώσουμε πληροφορίες που δεν είναι δημόσιες, θα μας το ζητούσαν άλλωστε αν ήταν δημόσιε οι πληροφορίες, κοινές πληροφορίε. έπρεπε να συντονιστούμε με τι δημόσιε αρχέ που ενδεχομένω είχαν τέτοιε πληροφορίε ή έχουν το νομικό δικαίωμα να αποκτήσουν τις πληροφορίες και το κάναμε αυτό ερχόμενοι σε επαφή με την αστυνομία της Μάλτας. Και έδωσε τελικά η αστυνομία της Μάλτας τις πληροφορίες που ζητούσε η Όλαφ. Αυτή ήταν η μόνη εμπλοκή της Υπηρεσίας Συντονισμού Καταπολέμησεως των Απατών στην όλη ε, έρευνα, αλλά εξελίχθηκαν τα πράγματα με τέτοιο τρόπο που δεν ενημερωθήκαμε για τα τεκτενόμενα στην έρευνα, όπως θα έπρεπε να γίνει, διότι από την άποψη της Επιτροπής Εποπτείας έπρεπε εγώ να βλέπω πώς δρά σε αυτές τις περιπτώσεις η Όλαφ. Βέβαια, πρόκειται ιδιαίτερη περίπτωση, διότι αφορά έναν ε, υψηλά ιστάμενο άνθρωπο, αλλά θα ανέμενα να ακολουθεί το πλήρως η διαδικασία. Και όσον αφορά αυτέ οι υπηρεσίε συντονισμού, το ΣΑΦΚΟ ακολουθήσαμε τι διαδικασίε. Όταν ελέγχουν οι συνάδελφοί μα του φακέλου αυτή τη υποθέσεω, συμπεραίνουν και συμπεραίνουμε ότι αυτή είναι η μόνη σχέση μεταξύ Όλαφ και ΑΦΚΟΣ Μάλτα, όσον αφορά αυτή την υπόθεση Νταλή. Πείτε μου λοιπόν τότε γιατί, θα μου πείτε γιατί αποσύρεστε από την υπόθεση Ντάλι και δεν περιμένα, δεν περίμενα τα μέσα ενημέρωση να μου πούν να παραιτηθώ. Παραιτήθηκα την επόμενη μέρα αμέσω, πριν μου πει κανεί τίποτα ότι πρέπει να αποσυρθείτε, να παραιτηθείτε. Το έκανα διότι είμαι υπήκο της Μάλτας. Θεωρώ ότι αν δεν είχα παραιτηθεί θα θεωρούσαν ότι κατά κάποιο τρόπο επηρέαζα την υπόθεση Νταλή, κάτι που δεν θέλω. Δεν θέλω να υπονομεύσω και να επηρεάσω οποιαδήποτε υπόθεση και εξήγησα στους συναδέλφους αυτό που σας εξήγησα εδώ, σε όλους σας. Τον μικρό ρόλο που έπρεπε να παίξουμε μέσω των διατάξεων περί διοικητικής συνεργασίας και είπα ότι για να φαίνεται ότι ήμασταν εξάρτητοι από την όλη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει η Εποπτική Επιτροπή και να μην να μην ε, επηρεάσουμε τι εξελίξει, διότι υπήρχαν πολλέ κατηγορίε. Ήξερα ότι οι συνάδελφοί μου είναι αρκετά ικανοί να χειριστούν την ε, υπόθεση και έχω κάθε πεποίθηση ότι με κάθε επαγγελματισμό θα εξετάσουν και θα χειριστούν αυτήν την υπόθεση. Ευχαριστώ πολύ. Εδώ από τα μέλη της Επιτροπής υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Όχι. Α, ο κύριος Γκάια ήθελε. Παρακαλώ. Όχι, δεν είναι ερώτηση. Α, όχι, είχα, έχω ακόμη μια ερώτηση. Ε, κοιτάξτε. Αν έχει κάποιος την εντύπωση ότι μεταξύ Προέδρου της ομάδας και ημού υπάρχουν καμία διαφορές, σε παρακαλώ πάρε αυτή την ανακοίνωση τύπου, βάλτε πάνω στο γραφείο σου και καρφίτσο την και κάρφωσέ την επάνω. Ο πρόεδρος της ομάδας μου μετά τις συζητήσεις με τον κύριο Κέστερ με ενημέρωσε και το θέμα νομίζω έχει διευκρινιστεί. Δεύτερον, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί να μην ε, αποφανθούμε με βάση την περίπτωση Ντάλι τι πάει καλά και τι πάει άσχημα με την Ντάλι. Το ξαναείπα και το λέω ακόμη. Δεν είμαστε δικαστήριο εδώ. Δεν είμαστε εμείς που θα πρέπει να αποφασίσουμε αν κάποιος είναι αθώος ή ένοχος σε τέτοιες περιπτώσεις. Ή όλα αυτά αποφασίζει αυτά. Και η Επιτροπή Εποπτείας της Όλαφ πρέπει να ασχολείται με τα δικαιώματα των κατηγορουμένων. Έτσι αντιλαμβάνομαι εγώ το ρόλο τους. Δεν είναι σαν τους ε, κριτές ε, στις, ε, γυμναστικές διοργανώσεις που θα πρέπει να σηκώνουν ένα νούμερο μετά από την επίδοση κάθε διαγωνιζομένου. Τώρα, εάν είναι επαρκείς οι δυνατότητες λειτουργίας της, επιπτω... Ε, της ε, Επιτροπής Εποπτείας της Όλαφ, βεβαίως να το συζητήσουμε. Υποστηρίζω βεβαίως αυτά τα οποία υπόθηκαν. Αλλά να μην μπλέκουμε πράγματα που δεν πρέπει να τα μπλέκουμε, γιατί αλλιώς είναι ολιστηρή η οδός Ίσως κάποιοι να νομίζουν ότι πρέπει να παίξουν τον Sherlock Holmes. Ίσως κάποιοι να θέλουν να πούνε ορισμένα πράγματα στους δημοσιογράφους. Αλλά δεν είναι αυτός ο ρόλος μας. Πρέπει να είμαστε πεπισμένοι ότι δεν υπάρχει κάποια παρατημία στην περίπτωση Ντάλι. Να μιλήσουμε για τον τρόπο λειτουργίας της Εποπτικής Επιτροπής της Όλαφ. Υποστηρίζω αυτά που υπόθηκαν προς αυτήν την κατεύθυνση. Νομίζω ότι κάναμε αυτά που είναι απαραίτητα. Και αν αισθάνονται ότι τους φημώνει ο κύριος Κέσλερ είναι όλοι σοβαρά και υπεύθυνα άτομα. Άκουσα τι είπαν τα μέλη της Επιτροπής. Ότι υπάρχουν ε, συνεχώς ε, διοικητικές ε, παρεμβάσεις και μικροσυγκρούσεις και ταλαιπωρίες. Αυτό να αντιμετωπιστεί βεβαίως. Αλλά να αφήσουμε την Εκκλησία στο μέσο του χωριού. Ωραία λέει ο Πρόεδρος. Υπάρχει πίεση χρόνου. Πιστεύω λοιπόν ότι θα έπρεπε να καταλήξουμε για το θέμα αυτό πριν δώσω το λόγο στη συνάδελφο Αγιάλα Σέντερ και μετά στην εισηγήτρια. Ως πρόεδρος όμως της Επιτροπής να διευκρινίσω τα εξή. Προτείνω να καλέσουμε τον κύριο Κέστλερ ενώπιόν μας. Συζητάμε ούτως ή άλλως συχνά με τον Γενικό Διευθυντή ναι, ναι, θα μιλήσετε κυρία Γκρέσλε και ο κύριος Μίλντερ. Εντάξει, θα υπάρξει μια περαιτέρω ανταλλαγή απόψεων. Προτείνω λοιπόν, κύριε Ντένουλφ και μέλη της Επιτροπής Εποπτείας, αυτά που ακούσαμε εδώ, να τα συζητήσουμε με τον κύριο Κέσλε, που είναι ο Γενικός Διευθυντής της Όλαφ. Ετέθησαν ορισμένα θέματα που πρέπει να τα εξετάσουμε. Συνοψίζοντας λοιπόν, προτείνω αυτό. Δεύτερον, οι περικοπές προσωπικού που μειώνουν τη δυνατότητα λειτουργίας μιας εποπτικής αρχής της οποίας τα μέλη μερικώς ασχολούνται με αυτόν τον ε, τομέα. Νομίζω ότι είναι λογικό αυτό. Και δεν είναι χωρίς σημασία αυτό το θέμα. Εφόσον, όπως ξέρετε, ο προπολογισμό της Ένωσης είναι 129 δις και εφόσον θέλουμε να υιοθετούμε και να ακολουθούμε αρχές κράτους δικαίου, πρέπει να υπόκειται σε έλεγχο και η Όλαφ και η Επιτροπή Εποπτείας είναι η αρμόδια να ελέγχει την Όλαφ. Και βεβαίως και η πρόσβαση στα κείμενα των υποθέσεων. Κοιτάξτε, μήπως ε, οι δύο θέσεις που σας αφαίρεσαν προσωπικού αυτή τη στιγμή ασχολούνται με το να διαγράφουν τμήματα των κειμένων που θα σας στείλουν. Καλά, αστεία τα λέω αυτά. Να δώσω τώρα το λόγο στους συναδέλφους ε, που, το, που ζήτησαν το λόγο. Πρώτος ο κύριος Μιούλντερ και μετά η συγγετρία, παρακαλώ. Όχι, πρώτη κυρία Σέντερ. Ασέντερ, ναι. Με συγχωρείτε, κράτησε πολύ ψηφοφορία στην Επιτροπή Μεταφορών για το πακέτο για τις ορομεταφορές, αλλά με ενδιαφέρει πάρα πολύ το θέμα αυτό και ευχαριστώ που μπόρεσα να έρθω για να θέσω ορισμένε ερωτήσει. Συμφωνώ με όλα όσα είπε ο κύριος Γκάιρος, συντονιστή μου, και κυρίω τονίζω ότι για μα η Επιτροπή Εποπτείας είναι οργανισμό κλειδί για να εγγυηθεί και να προστατεύσει την Όλαφ, να εγγυηθεί την ανεξαρτησία τη, για να αποφύγουμε ακριβώς να γίνονται λάθη ή να γίνονται ενέργειες προς τα μέσα μαζική ενημέρωση που να δημιουργούν καταστάσεις αρνητικές, όπως αυτή που είδαμε, όπου όλα τίθενται ένα αμφιβόλο. Σίγουρα η Επιτροπή Υποπτίας πρέπει να είναι σε θέση να προστατεύει την ανεξαρτησία της Όλαφ, να προστατεύει λοιπόν ένα ε, οργανισμό που ε, βεβαίως πρέπει να είναι ανεξάρτητη από την Κομισιόν, αλλά εξαρτάται από αυτήν και την ελέγχει παράλληλα. Στηρίζουμε λοιπόν το ρόλο της ε, Επιτροπής Εποπτείας και επίσης λαμβάνουμε πάρα πολύ τα δικαιώματα των ε, υποέρευνα. Βεβαίως πρέπει να υπάρχει διοντολογία, όπως είπε και η κυρία Γκρέσλε. Στόχος μας είναι να υπάρχει μεγαλύτερη εγγύηση των δικαιωμάτων αυτών γιατί αλλιώς θα είμαστε ευάλωτοι. Θέλω να σας ρωτήσω γιατί κάτι το οποίο δεν κατάλαβα. Ο κανονισμός λέει ότι εσείς έχετε δικαίωμα πρόσβασης στις έρευνες, ότι πρέπει λοιπόν με βάση τις έρευνες πρέπει να έχετε πρόσβαση, αλλά αναφερθήκατε σε μια συμφωνία εργασίας ότι δέχεστε να σας, να σας δίνουν μόνο μία συνόψιση των υποθέσεων. Μπορείτε να μας δώσετε αυτή την συμφωνία εργασίας για να δούμε τι είναι δυνατόν να απαιτήσουμε ή όχι. Γιατί δεν είναι δυνατόν εμείς να απαιτούμε να σας δώσουν όλη την τεκμηρίωση ενώ εσείς έχετε συμφωνήσει να σας δίνουν μόνο μια συνόψιση. Και συμφωνώ απόλυτα με το ότι το προσωπικό της Επιτροπής σας πρέπει να είναι επαρκής για να παίζετε ουσιαστικά τον ουσιώδη ρόλο σας για να εγγυηθείτε την εξαρτησία της Όλαφ και τα δικαιώματα των ερευνομένων και για να αποφεύγονται καταστάσεις όπως η σημερινή που αποδεικνύει ότι κάποια στιγμή έγιναν λάθη. Δεν είναι δυνατόν οι πολίτες να έχουν την εντύπωση ότι υπάρχει διαφθορά, πάτες, ότι δεν υπάρχει επαρκής εποπτεία Υποστηρίζω απόλυτα τα καθήκοντά σας, την εργασία σας. Πρέπει να βεβαιωθούμε ότι η συνεργασία, μας, η συνεργασία σας με την Όλαφ λειτουργεί σωστά. Και αν μπορείτε να ζητήσετε να σας δίνονται εκθέσεις. Ο κύριος Μιλντερ. Χαίρομαι που την επόμενη φορά θα καλέσουμε τον Γενικό Διευθυντή της Όλαφ να τον ρωτήσουμε να μας τα πει από τη δική του πλευρά. Καλό θα ήταν όμως να έχουμε και εκπρόσωπο της Επιτροπής Εποπτείας ταυτόχρονα για να ακούσουμε την ίδια ώρα τα επιχειρήματα των δύο μερών. Ωραία. Ευχαριστώ η κυρία Γκρέσλε. Δεν με πειράζει παρόλο που δεν το βρίσκω τόσο σημαντικό. Ας το δούμε. Το έχουμε συζητήσει το θέμα. Όχι την τελευταία φορά που ήταν και κλεισμένο των θυρών. Την πρώτη τελευταία φορά όμως του έθεσα το θέμα ακριβώς αυτό που μου είπατε εσείς. Και έγινε συζήτηση μαζί του. Και τον ακούσαμε τι είχε να πει. Γι' αυτό δεν είμαι αισιόδοξη και σας το λέω γιατί πραγματικά ο παχυδερμισμός αυτός ε, με ενοχλεί τρομερά. Δεν επιτρέπεται, έτσι είναι. Εν πάση περιπτώσει. Εντάξει. Εγώ συμφωνώ, όποτε θέλετε θα συνεργαστώ κι εγώ. Πάντως ε, το αποτέλεσμα πρέπει να είναι πιο συγκεκριμένο από την περασμένη φορά που τον είδαμε επί δύο ώρες. Επίσης, τα μέτρα λιτότητας δεν δικαιολογούνται παρόλο που μπορεί να θέλει κανείς να περικόψει στο προσωπικό. Γιατί πραγματικά βλέπω χιλιάδες, μόνο στην υπόθεση Ντάλι, χιλιάδες σελίδες ε, από τις ακροάσεις, από τις ανακρίσεις. Ε, είναι πολλή δουλειά. Για να δούμε λοιπόν τι θα αποφασίσει και η, η δικαιοσύνη στην Μάλτα. Ε, είναι γρήγορε οι διαδικασίε και οι εξελίξει τώρα. Νομίζω ότι σε κάθε περίπτωση που σα απασχολεί, που μας απασχολεί, ε, είναι μια ηλιδία λήθος για την αποτελεσματικότητα της δουλειάς της ε, Όλαφ. Είναι σημαντικό λοιπόν να βλέπουμε και μεμονωμένες υποθέσεις, γιατί ε, βεβαίως πρέπει να κάνουμε μια εξατομικευμένη προσέγγιση. Θα ήθελα να συζητήσουμε μετά και το τι θα κάνουμε με την υπόθεση Ντάλι που έχει τόσα ανοιχτά ερωτήματα ανεξάρτητα με την συνάντηση με εσά. Νομίζω ότι τον Ιανουάριο θα έπρεπε να ξανασυναντηθούμε για να μας πείτε για το αποτέλεσμα. Δεν ξέρω πότε θα ολοκληρωθούν οι έρευνες. Πάντως εμάς ε, μας είναι σημαντικό να ενημερωθούμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ τους συναδέλφους για την ε, ζωντανή αυτή συζήτηση και τέλος ε, έχετε το λόγο κύριε Ντανούφ για να απαντήσετε. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου που, για το γεγονός ότι μας ακούσατε. Τόνισα τη σημασία που έχει ο ρόλος της Επιτροπής της Εποπτικής κυρίως για το σεβασμό των ερευνητικών καθηκόντων της Όλαφ, που δεν έχει ελεγχθεί από άλλον παρά από την Επιτροπή Εποπτείας. Είναι σημαντικό αυτό. Αν συμφωνείτε και είμαι σίγουρος ότι συμφωνείτε, θα ήθελα να κλείσω αυτή την ακρόαση δηλώνοντας ότι θα σας στείλουμε μία επιστολή. Στην επιστολή θα ζητούμε την στήριξή σας επί των τεσσάρων σημείων που προανέφερα και εξήγησα και για να απαντήσω αυτό που είπε η Ισπανίδα εκπρόσωπος θα συμπεριλάβω και ένα αντίγραφο της συμφωνίας των τριών βημάτων που έχουμε, συμφωνίας που έχουμε με την Όλαφ για τη συνεργασία μας για την ώρα. Και αν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις και συνάδελφοί μου και εγώ είμαστε στη διάθεσή σας. Είμαστε στη διάθεσή σας, είσαστε πάντα ευπρόσδεκτοι στις ολομέλειές μας για διεξοδικότερη συζήτηση των θεμάτων που απασχολούν και εσάς και εμάς. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ντένολφ όλα τα, και όλα τα μέλη της Επιτροπής Εποπτείας. Πολύ καρποφόρα η ανταλλαγή απόψεων. Σας ευχαριστώ πολύ και προσβλέπουμε στην επόμενη συνάντησή μας. Σας ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, περνάμε στο επόμενο θέμα, το οποίο είναι το σημείο 7. Η επίσκεψή μας στην Λιθουανία για την οριστική πάυση λειτουργίας του πυρηνικού σταθμού Ιγναλίνα. Το συζητήσαμε αναλυτικά εδώ μας ζητήθηκε συμπληρωματική πληροφόρηση. Υποβλήθηκε από την Κομισιόν. Συμπεριλήφθηκε στην έκθεσή μας. Οπότε, να ευχαριστήσω για την παρουσία του τον ε, μόνιμο, εκπρόσωπο, μόνιμο αντιπρόσωπο της Λιθουανίας στο Κορεπέρα 1, Αρούνας Βιντσιούνας. ο οποίος μας παρακάλεσε να μας παρουσιάσει την άποψη της λιθουανικής κυβέρνησης Βεβαίως. Να τον ακούσουμε και μετά να ενημερωθούμε για την έκθεση. Καλώς ήρθατε. Παρακαλώ ε, ενημερώστε μας όπως ε, επιθυμείτε συντόμως για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για συγκεκριμένα μέλη του Κοινοβουλίου. Εκτιμώ πράγματι τη δυνατότητα που έχω να μιλήσω στην Επιτροπή σε σημαντικότατο αυτό θέμα για τη Λιθουανία, για τον πυρηνικό σταθμό, τον παροπλισμό του Ιγναλίνα. Εμεί κλείσαμε αντιδραστήρε όπω συμφωνήσαμε στην ταξιακή μα συμφωνία 2004-2009 και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφώνησε να βοηθήσει σε αυτό το τεράστιο καθήκον για τον παροπλισμό των πυρηνικών αυτών αντιδραστήρων. Λοιπόν, είναι η πρώτη φορά στην ιστορία που γίνεται ε, παροπλισμός τέτοιου μεγέθους αντιδραστήρων και τέτοιου είδους αντιδραστήρων. Ε, χρειάστηκε να... Δεν υπήρξε παρέκκληση από τους κανόνες. Αυτό αναφέρεται και στην έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου. Η διαδικασία παροπλισμού του σταθμού έχει δρομολογηθεί και έχει κλείσει και ο δεύτερο αντιδραστήρα εδώ και δυόμιση χρόνια μόλι. Και η χρήση των πόρων σε σχέση με τα αποτελέσματα ε, μα δείχνει ότι τα πράγματα είναι ικανοποιητικά. Με ένα συμβαλόμενο μέρο έχουμε πρόβλημα. Ε, με το μόνο που ήρθε εδώ στην Επιτροπή και δεν είναι προβλήματα γραφειοκρατικά. Ως το θέμα τη πυρηνική ασφάλεια είναι το πρόβλημα. Πριν από μερικέ μέρε αυτό ο ανάδοχο ζήτησε από ρωσική εταιρεία να κάνει εργασία στην Ιγναλίνα και αυτή είναι... Και είχαμε πρόσφατα εμπειρία ότι υπήρξε ένα σοβαρό πυρηνικό ατύχημα στην Ρωσία σε πυρηνικό αντιδραστήρα που κατασκευάσατε. Δεν μιλάμε τώρα για γραφειοκρατικό άχθο. Υπάρχει σοβαρό θέμα πυρηνική ασφάλειας και είναι κάτι στο οποίο δεν συμβιβαζόμαστε. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, οι αδίποτε νέα συμπεράσματα του ελεκτικού συνεδρίου και αν ε, παγώσουν οι, τελικά οι χρηματοδοτήσεις, έτσι υπονομεύεται η πυρηνική ασφάλεια. Και αυτή η απόφαση πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ ατυχής, δηλαδή αν μειωθούν τα κονδύλια. Παγώσουν μάλλον οι χρηματοδοτήσεις. Ευχαριστώ κύριε Μπρέσλερ για τη δήλωσή σας. Να επιστήσω την προσοχή των μελών στα συμπεράσματα της αντιπροσωπείας αυτά και να έχουμε υπόψη μας το χρονοδιάγραμμα. Πότε πήγαμε στην ε, μονάδα παραγωγής της Ινιαλίνα και αυτό που αναφέρατε είναι μόνο ένα κομμάτι των σύμπερα. Ήταν μόνο ένα μέλος αντιπροσωπείας. Θα δώσω τώρα το λόγο, ε, τον λόγο και στα άλλα μέλη, στον συνάδελφο Μπαλτσίτης. Ευχαριστώ συνάδελφοι. Καταρχάς, να ευχαριστήσω όλη την ε, αντιπροσωπεία ε, της Κοκομπή η οποία κατά την άποψή μου διαδραμάτισε έναν ιστορικό ρόλο σε 12 χρόνια υπήρξε σειρά ανεπίλητων προβλημάτων και με τη βοήθεια της επίσκεψης της αντιπροσωπείας ε, συζητούμε τα προβλήματα ε, εκτενώς όμως ε, δεν μπορώ να συμφωνήσω με τα συμπεράσματα της αντιπροσωπείας μετά από την επίσκεψη στο πυρηνικό σταθμό της Ιγναλίνα διότι ε, κατά την άποψή μου στο όλο αυτό θέμα στην όλη κατάσταση την περιπλοκότατη η κατανομή των ρόλων και η διανομή των ευθυνών ε, δεν έγινα με δίκαιο τρόπο. Πρώτα απ' όλα ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πρέπει να αναφερθεί. Από την απάντηση που δόθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατανοούμε σαφώς ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, μαζί με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανάπτυξη Ανοικοδόμηση είναι υπεύθυνη για την ε, εφαρμογή, για την υλοποίηση της οικονομικής βοηθείας που χορηγεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα συμπεράσματα δηλώνουν ότι καθυστερούν οι ε, υλοποίησεις κάποιων προγραμμάτων, κάποιων έργων που συνεπάγεται και αυξανόμενο κόστος όμως δεν συμφωνούμε ότι η Λιθουανία είναι η μόνη που φταίει για τις καθυστερήσεις. Το 2001 υπεγράφει συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Τράπεζας ε, Νικόδημης και, και της Λιθουανίας που και αναφέρει σαφείς κανόνες που πρέπει να πληρούνται για την υλοποίηση των έργων, έγκαιρη υλοποίηση των έργων. Σύμφωνα με τη συμφωνία, μία ομάδα ε, διαχείρισης του έργου πρέπει να συσταθεί και μία μεικτή επιτροπή αυτή η ομάδα κοινή διαχείρισης συστάθηκε, ήταν αρκετά ενεργή στην αρχή. 26 εμπειρογνώμενες συμμετείχαν. Η διαδικασία επιλογής παρακολουθεί το πολύ σαφώς από την Ευρωπαϊκή Τάπεζα ε, Ανοικοδόμησης και Ανάπτυξης. Ε, αλλά η ε, ομάδα όμως διαχείρισης μειώθηκε σε μέλη. Έχουμε μόνο 6 εμπειρογνώμονες βασικός τους ρόλος ήταν να επιλύουν προβλήματα όταν αυτά ανακύπτουν και θα ήθελα να ενημερώσω τα μέλη της Επιτροπής λέγοντας ότι η ομάδα διαχειρίσεως των έργων ε, έλαβε τέσσερα 43 εκατομμύρια για τα έργα. Ε, έγινε συνέλευση των δωρητών και δύο φορές το χρόνο έπρεπε να τους ενημερώνει η Λιθουανία για την υλοποίηση των έργων, όμως δεν είχαμε κάποια αντίδραση. Μόνο μετά την επίσκεψη της Επιτροπής, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε να θέτει τα προβλήματα των διαφόρων καθυστερήσεων. Σα επιστώ λοιπόν την προσοχή επί του γεγονότος ότι η Λιθουανία δεν κινείται μόνη της. Έχουμε και άλλα τρία μέρη. Έχουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα για, για την Ανάπτυξη, και ε, την ανάδοχο εταιρεία, την Newcam, η οποία διαπραγματεύτηκε κάποιους όρους με την ε, τράπεζα για το κλείσιμο, για τον παροπλισμό του εργοστασίου. Μετά για την πυρηνική ασφάλεια, συμφωνώ με τον κύριο Πρέσβη που εξέφρασε ανησυχίες όσον αφορά την πυρηνική ασφάλεια και νομίζω ότι είναι προς όφελος της Λιθουανίας και των άλλων χωρών προς συμφέρον τους να ε, υλοποιούνται να εκτελούνται τα καθήκοντα των αρμοδίων φορέων με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Δεν πρέπει να υλοποιούνται έργα και εργασίες που δημιουργούν αμφιβολίες και ίσως να μειώνει το επίπεδο της πυρηνικής ασφάλειας. Άρα η απέτηση της Λιθουανίας να δοθούν έγγραφα ε, όσον αφορά τα έργα είναι κάτι δικαιολογημένο και δεν μπορεί να θεωρηθεί αυτό σαν μοναδικός αποκλειστικός λόγος για τις καθυστερήσεις των έργων και ε, για τη μη τήρηση των προθεσμιών. Το 2017 είναι η τελική προθεσμία. Πρέπει να πω ότι το πρωτόκολλο 4 της Συμφωνίας Ένταξης αναφέρει ότι χώρες όπως, αυτές οι χώρες όπως είναι η Λιθουανία ε, πρέπει να σηκώσουν ένα τρομερό οικονομικό βάρος που απορρέει από τον παροπλισμό μέσα στις εγκατάστασεις και δεν μπορεί μια χώρα μόνη να χρηματοδοτήσει τα πετούμενα έργα. Η πρόταση λοιπόν η οποία υπευλήθη και τα συμπεράσματα της αντιπροσωπείας που αφορούν την προθεσμία του 2017 δεν ταιριάζουν με τις απαιτήσει του πρωτοκόλου και τις διατάξεις του πρωτοκόλου. Αυτό κατά την άποψή μου δείχνει έλλειψη σεβασμού της συμφωνίας ένταξης και αυτό μπορούν να το εξετάσουν και να αποφανθούν ε, νομικοί εμπειρογνώμονες. Η επίσκεψη νομίζω ήταν πάρα πολύ θετική εξέλιξη. Συμφωνώ ότι πρέπει να επιληθεί το πρόβλημα. Θα πρέπει να βρεθεί μια πιο δίκαιη λύση, ούτω ώστε να βρούμε έναν τρόπο ούτω ώστε να λειτουργούν αποτελεσματικά όλοι οι θεσμοί και έγκαιρα. Αυτό θα είναι καλή εμπειρία για άλλα προγράμματα αφοπλισμού παρομοίων εγκαταστάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και νομίζω ότι τα συμπεράσματα της Επιτροπής θα πρέπει να τροποποιηθούν, να διορθωθούν, ούτω ώστε να μπορούμε να συμβάλλουμε στην επίλυση τέτοιων προβλημάτων, όχι μόνο στη Λιθουανία, αλλά οπουδήποτε αλλού, σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Ε, first Καταρχάς, να υπογραμμίσω ότι όλα τα μέλη της αντιπροσωπείας κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η πυρηνική ασφάλεια είναι το πρώτο στο μέλημά μας. Αυτή είναι η πρώτη, είναι το πρώτο πόρισμα. Δεύτερον, προβλέπεται πολύ μεγάλο ποσό στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, 1,367 δις ευρώ τόσο θα δαπανίσει η Ένωση για να παροπλιστεί ο σταθμός Ιγναλίνα. Στην έκθεση επίσης αναφέρεται και η πρόοδος που έχει σημειωθεί, αλλά και τα προβλήματα που έχουν ανακύψει. Δεν λέει η έκθεσή μας πουθενά ότι η κυβέρνηση της Λουφανίας είναι αποκλειστικά υπεύθυνη. Αν κοιτάξετε, θα δείτε ότι είναι ιδιαίτερα αντικειμενική και είναι η έκθεση αυτή πόρισμα όλης της αντιπροσωπείας μας. Πρέπει να εμείνουμε στη γραμμή μας, συνάδελφε Μπαλτσίτη. Όλοι όσοι συμμετέχουν πρέπει να συνεργαστούν για να εξευρεθούν λύση, λύσεις. Και νομίζω ότι είναι λυπηρό το ότι κάποιοι αρμόδιοι ή ίσως ε, κάποια μέσα μαζικής ενημέρωσης ανέφεραν μονομερώς τα πορίσματα της ε, επίσκεψής μας. Δεν ξέρω τώρα γιατί. Αλλά εμείς υιοθετήσαμε αντικειμενικά συμπεράσματα και πρέπει να εμείνουμε σε αυτά. Στο παρελθόν δεν ψηφίζουμε για τις εκθέσεις αντιπροσωπιών, δεν ψηφίζαμε, αλλά σας υπενθυμίζω ότι αμέσως μετά την επίσκεψη στη Λιθουανία, πριν από τρεις μήνες, υιοθετήσαμε αυτό το πόρισμα και θα πρότεινα να επιμείνουμε σε αυτά που είχαμε συμφωνήσει τότε. Θέλει κανείς το λόγο. Η κυρία Γκρέσλε. Συμφωνώ. Αυτά ήταν τα πορίσματά μας. Αυτά είναι και σήμερα αλλά έχουμε εδώ και την Επιτροπή. Θα ήταν ε, καλό να λάβουμε μια ενημέρωση. Έχουν περάσει τρεις μήνες. Πιστεύω ότι είναι σκόπιμο να τους ακούσουμε. Πρόεδρος, ίσως ε, μετά την επίσκεψή μας να έχουν επιληθεί όλα τα προβλήματα. Ρωτάω λοιπόν την Επιτροπή. Μπορείτε να μας πείτε ότι έληξε ο συναγερμός. Έχει σημειωθεί πρόοδος τους τελευταίους τρεις μήνες. Παρακαλώ, σε ποιον να δώσω το λόγο. Η κυρία Πλομχίβο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Να σας ενημερώσω. Καταρχήν, μας ενδιαφέρει πολύ η έκθεσή σας και την παρακολουθούμε από κοντά. Η Κομισιόν συμφωνεί ότι το κλείσιμο του αντιδραστήρα 2 είναι η πρώτη προτεραιότητα. Δεν μπορώ να σας πω ότι όλα πάνε πρίμα. Στην τελευταία συνέλευση των συμμετεχόντων είπαμε ότι τα δύο μέρη, από τη μία πλευρά δηλαδή η υπεύθυνη για το πυρηνικό εργοστάσιο και την άλλη ο ανάδοχος, θα καταρτήσουν οδικό χάρτη και το έκαναν. Όμως, ακόμα και που έγινε ο οδικός χάρτης, δεν μπορούσαν μετά να υποβάλουν κοινή έκθεση που αυτό όμω είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει κοινή έκθεση που θα αποδεικνύει ότι τα δύο μέρη συμφωνούν για την υλοποίηση, γιατί μόνο στα χαρτιά δεν φτάνει. Δυστυχώ, λοιπόν η κατάσταση για μα είναι απαράδεκτη. Για το β δεν βλέπουμε πρόοδο στην πραγματική υλοποίηση. Και τι είναι αυτό, ότι θα πρέπει να παροπληστεί ο δεύτερο αντιδραστήρα, θα έχουμε λειτουργικότητα και δεν θα έχουμε κίνδυνο ασφάλεια. Συμφωνούμε λοιπόν με την Λιθουανική Αντιπροσωπεία και την έκθεσή σας ότι δεν μπορεί να γίνονται συμβιβασμοί σε θέματα ασφάλειας. Τα λαμβάνουμε αυτά υπόψη. Θα, θα συναντηθούν πάλι το Δεκέμβριο τα συμμετέχοντα μέρη και θα πιέσουμε ε, για, όσο μπορούμε για να επιτευχθεί, να βοηθήσουμε να υπάρξει πρόοδος. Επίσης, ε, μπορεί η συνέλευση να καταλήξει σε αυτό που αναφέρθηκε τον Ιούνιο, να, να, δηλαδή να υπάρξει αναστολή της συμφωνίας που καλύπτει το Β1, δηλαδή την ενδιάμεση αποθήκευση και την, ε, ε, ε τον και ε, μπορεί αυτό να σημάνει το τέλος της συμφωνίας. Και δεν θα μπορεί η Λιθουανία ε, μαζί με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότηση και Ανάπτυξη να λύσουν το θέμα. Τώρα εκεί που διαφοροποιείται η Κομισιόν είναι στο πλήρε πάγωμα. Πάλι συμμεριζόμαστε τη δήλωση του πρέσβη ότι ε, υπήρξε πρόοδος στον, στη διάλυση, τον παραπλησμό και γι' αυτό διετέθησαν σωστά και αποτελεσματικά και αποδοτικά τα κονδύλια. Η Κομισιόν εδώ προτείνει αναστολή μόνο. Είναι εναλλακτική. Δεν αποφασίσαμε οριστικά, αλλά είναι μια εναλλακτική που θα συζητηθεί στην επόμενη συνέλευση ούτως ώστε αυτή η συμφωνία ε, για το B1 να ανασταλεί. Έχουμε την πρόθεση όμως να συνεχίσουμε να χρηματοδοτούμε τα άλλα έργα, γιατί εκεί υπάρχει σαφής πρόοδος. Χωρίς όμως να εφαρμοστεί το έργο Β1, υπονομεύεται ολόκληρη διαδικασία. Αυτό είναι αλήθεια. Και με αυτή την ευκαιρία να πω ότι η Κομισιόν ε, έχει επισημάνει τις, τις καθυστερήσεις εδώ και καιρό, μας ανησυχούν και ψάχνουμε να βρούμε διαφορετικούς τρόπους για να λύσουμε το θέμα. Και η Κομισιόν έκανε πολλές προσπάθειες και αφιέρωσε και ανθρώπινους πόρους σε αυτά τα έργα. Πήγαμε σε συναντήσει για να διευκολύνουμε τη συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών μετά από αίτημα τη Λιθουανίας, ελπίζοντας ότι θα επιτελεί το πρόοδο. Αλλά είμαστε τώρα σε μια κατάσταση που τη θεωρούμε πλέον απαράδεκτη. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Πολύ σημαντικές οι πληροφορίες σας. Να ρωτήσω και κάτι ακόμη ως συμπέρασμα της ε, επίσκεψης της αντιπροσωπείας μας, εμείς μεταξύ άλλων καταλήξαμε ότι πρέπει να υπάρχει μια επιτροπή κοινή μεταξύ της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και της Λιθουανίας για να διευκολύνει ανταλλαγές πληροφοριών. Ή, συμφωνούμε εδώ με τον ε, συνάδελφο Μπαλτσίδης και όλοι οι άλλοι συνάδελφοι επίσης, ότι το βασικό μας μέλημα και κύριε Πρέσβη, θα ήθελα να το πω αυτό και για τη λιθουανική κυβέρνηση. Το βασικό μέλημα λοιπόν για μας είναι ότι οι μελλοντικέ συγκρούσεις που συνηθίζονται σε ένα τέτοιο μεγάλο έργο θα πρέπει να βρίσκονται μέσα σε ένα πλαίσιο ε, μηχανισμού επίλυσης διαφορών. Το έργο αυτό θα πρέπει να ολοκληρωθεί το ταχύτερο δυνατόν προς το συμφέρον του λαού, αλλά και για λόγους πυρηνικής ασφάλειας. Αυτές είναι οι δύο βασικές συνιστώσεις. Να είμαστε αποτελεσματικοί και αποδοτικοί ε, σε σχέση με την πυρηνική ασφάλεια και λαμβάνοντας υπόψη και τους δημοσιονομικούς μας στόχους. Ίσως η Κομισιόν μπορεί να μας ενημερώσει σχετικά με την σύσταση αυτή, αυτής της Επιτροπής έχει γίνει ήδη. Πώς κρίνεται δηλαδή αυτό το θέμα ενός μηχανισμού επίλυσης διαφορών. Υπάρχει επιτροπή, δεν είναι επιτροπή EBRD Λιθουανίας, είναι κοινή επιτροπή καθοδήγησης και υπάρχει εδώ και κάποια χρόνια και συμμετέχει και η Κομισιόν. Και υπήρχε επανειλημμένο αίτημα από τη Λιθουανική κυβέρνηση σε όλες αυτές τις συναντήσεις να συμμετέχει η Κομισιόν και ανταποκρίθηκε η Κομισιόν στο αίτημα αυτό. Και σε ε, όλες τις ρυθμίσεις είμαστε, ενώ παλιότερα όχι. Και κατάλαβα ότι οι Λιθουανοί το εκτίμησαν πάρα πολύ αυτό. Και δεν ε, βλέπουμε, δεν βλέπουμε δηλαδή να εξευρίσκεται η λύση αν η Λιθουανία συναντάται μόνο με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης ο κύριος ε, Μπαλτσίτης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εκτιμούμε πάρα πολύ ε, την συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά τα θέματα πυρηνικής ασφάλειας και όσον αφορά πολλές άλλες πτυχές. Και εγώ, κύριε Πρόεδρε, είμαι ένας άνθρωπος που συμβιβάζεται Πάντα προσπαθώ να επιτυγχάνω συμβιβασμούς. Κρίνοντας από αυτά που μόλις ακούσαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μπορούμε να πούμε ότι έχει επιτευχθεί κάποια πρόοδος και από τις δύο πλευρές και θα επαναλάβω εκ νέου ότι αυτό είναι το αποτέλεσμα του έργου της Επιτροπής Ελέγχου Προϋπολογισμού και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Ίσως θα μπορούσαμε να επιδιώξουμε συμβιβασμό στη διατύπωση της τελευταίας φράσης που αναφέρεται στην πάυση της χρηματοδότησης για τον παροπλισμό το 2017. Εάν συμφωνήσουμε επ' αυτού, τότε όλες οι πλευρές θα ικανοποιηθούν και θα έχουμε μια πολύ καλύτερη απόφαση που θα ληφθεί σε πολιτικό επίπεδο. Σας ευχαριστώ. Äh, η κυρία Γκρέσλε. Εάν εξαρτιόταν από μένα θα έκλαινε ήδη το 2014. Με συγχωρείτε, δεν μπορώ να συμφωνήσω αλλαγή. Εάν επεκταθεί, είχε θελούσιους, θελουσίως πει η Ένωση ότι μπορούσε να επεκταθεί. Με συγχωρείτε, όμως εγώ δεν συμφωνώ. Όχι, δεν συμφωνώ. Πρόεδρος. Τώρα, πώς να επιλύσουμε αυτή τη διαφορά. Να συνοψίσω τη έκθεση και μετά την ε, δήλωση της Επιτροπής θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε να αλλάξουμε τη διατύπωση από εκεί που λέει να παγώσει, να βάλουμε να ανασταλεί. Αυτό θα ήταν δυνατό. Γιατί όχι? Γκρέσλερ. Συμφωνώ. Κοιτάξτε, κοιτάξτε, καλύτερα. Εάν ε, δεχθούμε κάτι περισσότερο, στην ουσία τα παρατάμε. Με συγχωρείτε, είμαι κατά του να υποχωρήσουμε στο σημείο αυτό. Γιατί έχω την εντύπωση ότι μέχρι τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με μικρά βήματα κάτι επέτυχε. Δεν συμφωνώ να αλλάξουμε τα πορίσματα στα οποία είχαμε όλοι καταλήξει και πολλοί λείπουν τώρα. Να εμείνουμε λοιπόν και η Κομισιόν που έχει τη δική της ευθύνη μπορεί να λάβει άλλες αποφάσεις αν θέλει και θα τα ξαναπούμε μετά σε δύο μήνες. Θα ελέγξουμε τι επετεύχθη. Ο Γένς, νομίζω, κάλεσε τον αρμόδιο επίτροπο. Εγώ δυστυχώς δεν θα μπορέσω να παρευρεθώ γιατί πρέπει να πάω σε μια κηδεία στην περιοχή μου. Αλλά νομίζω ότι θα έπρεπε να μείνουμε στην παρούσα διατύπωση. Okay. Um... Ποιος άλλος? Ο κ. Μπαλτσίτης. Ευχαριστώ. Η κυρία Γκρόσλε ανέφερε ότι όλα συμφωνήθηκαν. Με συγχωρείτε, εγώ δεν θυμάμαι. Να με ρώτησε κανείς αν συμφωνώ εμένα για το θέμα αυτό. Όλοι έχουμε προσωπικές απόψεις για πολλά θέματα. Αλλά, σε τελευταία ανάλυση, συζητάμε για υποχρεώσεις, δεσμεύσεις Οπότε νομίζω ότι εμείς εδώ ως Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού αυτό ισχύει και για άλλες επιτροπές θα μπορούσαμε να βρούμε μια διέξοδο από αυτή την κατάσταση τροποποιώντας ελαφρώς το κείμενο. Μπορούμε να αναφερθούμε σε υποχρεώσεις της Ένωσης το έχουμε ήδη αναφέρει επανειλημμένα σε προηγούμενες περιπτώσεις και ευχαριστώ. Από την άποψή μου, δεν απέχουν και τόσο πολύ οι δύο απόψεις που ακούστηκαν. Να σας υπενθυμίσω ποιο είναι το πλαίσιο λειτουργίας της Επιτροπής μας. Στόχος μας πρέπει να είναι να δαπανώνται όσο το δυνατόν λιγότεροι πόροι. Τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν. Δεν μπορούμε να αποδεχθούμε ο ανάδοχος, κάποια άλλη φορείς κάποιοι εργοδότες εάν δεν κάνουν αυτά που πρέπει και αυτά που είναι στο χέρι τους για να λήξει η διαδικασία και να λυθεί το πρόβλημα ώστε να τον πιο σύντομα, αυτό δεν μπορούμε να το δεχτούμε. Πρέπει να εμείνουμε λοιπόν σε αυτά που λέει αυτή η κουκίδα στην ε, σελίδα 7 ότι πρέπει να εμείνουμε σε αυτά που λέγεται ότι πρέπει να ανασταλούν και να παγώσουν οι πληρωμές συγγνώμη, να συμφωνήσουμε στο να ανασταλούν μέχρι να υπάρξουν οι σχετικές ενέργειες μέχρι να υπάρξει ένας μηχανισμός για επίλυση διενέξεων. Υπενθυμίζω σε όλους ότι υπάρχει μια κοινή επιτροπή, μάλλον προτάθηκε από λιθουανική πλευρά, από το Λιθουανικό Ελεκτικό Συνέδριο, μια κοινή επιτροπή Ευρωπαϊκής Τράπεζας ε, Ανοικοδόμης Ανάπτυξης και Λιθουανίας. Και υιοθετήσαμε αυτή την πολύ λογική πρόταση από την λιθουανική πλευρά. Και έκτοτε υποστηρίζουμε αυτή την πολύ λογική πρόταση να περάσω τώρα στην τελευταία κουκίδα. Ξέρω, συνάλφε Μπαλτσίτης, ότι η λουθουμανική κυβέρνηση έδρασε με τρόπο κάπως ε, περιοριστικό και κατά τη γνώμη μου και λιγάκι αγενή. Τότε που καθόμαστε σε αυτό το περίφημο μέγαρο, ε, η ατμόσφαιρα κατά τη γνώμη μου ήταν λίγο περίεργη. Η λιθουανική κυβέρνηση ζητάει περισσότερα χρήματα και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Ωραία. Ωραία. Ας το διαπραγματευτούν στα πλαίσια του πολιετούς δημοσιονομικού προγράμματος, των πολιετών δημοσιονομικών προοπτικών. Αλλά εμείς και η γραμματεία που ήταν μαζί μου και εγώ ως πρόεδρος βρήκαμε αυτή την αρκετά ανοιχτή διατύπωση. Υπάρχει πρόταση από πλευρά τη ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Επιτροπή, που είναι η εκτελεστική αρχή μα, αντιμετωπίζει το θέμα αυτό. Εμεί είμαστε νομοθετικό σώμα. Διαβάζω λοιπόν την πρόταση. Η αντιπροσωπεία υποστηρίζει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αποδοθούν επιπλέον 230 εκατομμύρια για το 2014-2017 σε αυτή τη φάση θα πρέπει να τελειώσει η οικονομική στήριξη. Οποιαδήποτε νέα χρηματοδότηση στα πλαίσια των πολιτών δημοσιονομικών προοπτικών θα πρέπει να μπουν στο αποθεματικό μέχρι να υπάρξει πλήρης αιρεσιμότητα στα πλαίσια της αναθεώρησης του κανονισμού και να εγγυηθούμε την πλήρη αποτελεσματική χρήση των πόρων. Έτσι θα βοηθήσουμε να επιληθεί αποτελεσματικά το πρόβλημα. Αυτό μας ενδιαφέρει. Ποιος μπορεί να λύσει το πρόβλημα, όχι η Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού βεβαίω, σίγουρα. Όλοι οι άλλοι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Τράπεζα, η Ιγναλίνα, οι ανάδοχοι, δεν είναι στα χέρια μας. Εμείς κάνουμε μια έκκληση, καλούμε όλους τους εμπλεκομένους φορείς να μην συνεχίσουν να ε, διαπληκτίζονται, αλλά να επιχειρήσουν να υπάρξει μια επίλυση. Και τι δυνατότητε έχουμε για να πιέσουμε. Μόνο τον προπολογισμό. Για να πιέσουμε όλους τους εμπλεκομένους να επανέλθουν στην τράπεζα των πραγματεύσεων για να λύσουν το πρόβλημα. Πρέπει λοιπόν να εμείνουμε στο πόρισμα τη αντιπροσωπείας μας. Εάν τώρα κάποιοι προτείνουν άλλε διατυπώσει που μας διευκολύνουν όλου, εγώ βεβαίω να τι εξετάσω. Ω Επιτροπή πρέπει να δρούμε ενιαία, διότι Όλοι έχουμε τους ίδιους στόχους για το θέμα αυτό. Όλοι θέλουμε να εξοικονομήσουμε πόρους. Συνάδελφε Μπαλτσίτης. Κύριε Πρόεδρε, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Ο βασικός μας και γενικότερος στόχος είναι η επιτάχυνση της διαδικασίας και η αποτελεσματική χρήση των πόρων. Με τον παροπλισμό της Ιγναλίνας. Ο βασικός στόχο ήταν η πυρηνική ασφάλεια βέβαια. Σύμφωνο με όλα λοιπόν. Αν αφορούσαν μόνο την απορρόφηση των, των ε, κονδυλίων της Ένωσης. Υπάρχει όμως και ένα άλλο πρόβλημα. Η περίοδος μετά το 2017 Ίσως εκεί μπορούμε να βρούμε μια άλλη διατύπωση που θα λέει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε να αναλύσει την κατάσταση στο μέλλον και τα τρία μέρη ίσως θα μπορούσαν από κοινού να καθίσουν και να βρουν μια πιο ξεκάθαρη λύση, αλλά θεωρώ ότι αυτή η αυστηρή προϋπόθεση ότι θα πρέπει να σταματήσει η χρηματοδότηση το 2017 δεν συμφωνεί, με, δεν συνάδει με το γενικό στόχο της αναβάθμισης της ασφάλειας στην περιοχή. Γι' αυτό διαφοροποιούμε με τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής. Συγγνώμη, αλλά απευθύνω έκκληση να βρεθεί μια συμβιβαστική λύση εδώ. Μάλιστα. Ποιοι συνάδελφοι ζητούν ακόμη το λόγο. Είδα τον κύριο Μαρινέσκου που είναι και εισηγητής. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Δεν ήμουν στην αντιπροσωπεία αλλά επεσκέφθη την Ιγναλίνα πριν από αρκετούς μήνες, πάνω από 1,5 χρόνο συγκεκριμένα, διάβασα πολύ προσεκτικά την έκθεση και με έκπληξη είδα ότι δεν σημειώθηκε πρόοδος στις δραστηριότητες για τον παροπλισμό. Είδα ότι η κατάσταση έχει μείνει στα ίδια όπως πριν από 1,5 χρόνο και αυτό δεν εξυπηρετεί βέβαια την ασφάλεια και των πολιτών σας και της Ευρώπης γενικότερα. Συμφωνώ λοιπόν με τα συμπεράσματα της αντιπροσωπείας και όπως ξέρετε υπάρχει ένας κανονισμός βάσει του MFF, του Πολιτούς Δημοσιονομικού Πλαισίου, που αφορά την κατανομή των κονδυλίων για τις μελλοντικές δημοσιονομικές χρήσεις 2014-2020 για την περίοδο αυτή και εκεί προτείνει η Κομισιόν να είναι αυτή η τελευταία περίοδος χρηματοδότησης και των τριών πυρηνικών εργοστασίων και των τριών έργων σε αυτά. Και νομίζω ότι αυτή η πρόταση είναι πολύ σοφή. Προτείνεται δεν να κατανέμονται τα κονδύλια μόνο με βάση ενός σαφέστατου προγράμματος με πολύ ξεκάθαρες δραστηριότητες, με προϋποθέσεις και χρηματοδότηση παράλληλα. Και θα πρέπει να αναφέρεται και η πηγή της χρηματοδότησης. Γιατί το να στηρίζουμε τις συζητήσεις μόνο στην ασαφή διατύπωση της συνθήκης ένταξης ε, δεν είναι σωστό εδώ στο Κοινοβούλιο να το κάνουμε αυτό. Πρέπει να σκεφτούμε πώς θα λυθεί το πρόβλημα. Παράλληλα όμως θα πρέπει να εξοικονομούμε και χρήματα στην Ευρώπη. Εύκολα ζητάει κανείς χρήματα. Η σωστή δαπάνη των χρημάτων είναι πιο δύσκολο πράγμα. Γιατί όλα τα έργα διαθέτουν χρήματα για να δαπανίσουν από τον τωρινό, από την τωρινή κατανομή, <laughs> για να μην μιλήσουμε για το, τις μελλοντικές κατανομές, και δαπανούν πολλά ζητήθηκαν πολλά χρήματα για την ενέργεια γενικότερα. Ζητήθηκαν ε, στα πλαίσια της ε, ένταξης, όχι για τον, παρα, Τώρα θα πρέπει να δούμε με διαφορετικό μάτι αυτή τη δραστηριότητα. Είναι σωστή, είναι δικαίωμα βεβαίως του κράτους μέλους να ζητήσει χρηματοδότηση, γιατί αυτό προβλέπεται στη συνθήκη ε, προσχώρησης αλλά δεν λέει εκεί πουθενά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να χρηματοδοτεί τις δραστηριότητες κατά 100%. Συμπεραίνοντας λοιπόν, νομίζω ότι τα πορίσματα της αντιπροσωπείας πιστεύω ότι είναι καλά, σωστά και θα πρέπει να τα εγκρίνουμε κι εμείς. Να μην τροποποιήσουμε αυτά τα συμπεράσματα. Δεν θέλω να ξαναζητήσω το λόγο, γι' αυτό λέω, θέλω να μάθω. Τι προβλέπετε για την έκθεση που έχω αναλάβει στην Επιτροπή, γιατί πρώτη φορά είμαι σε αυτή την κατάσταση. Η έκθεση σταμάτησε. Στο τελικό της στάδιο, γιατί είχαν κατατεθεί τροπολογίες και σταμάτησε, αδικαιολόγητα πιστεύω εγώ, τέλο πάντων έγινε αυτό το πράγμα. Τώρα πήγε και επισκέφθηκε αντιπροσωπεία ε, την Ιγναλίνα και θέλω να μου πείτε τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Θα δοθεί νέα προθεσμία κατάθεση τροπολογιών. Θέλω να ξέρω επίσης πότε θα ψηφιστεί η έκθεση αυτή. Ευχαριστώ πολύ αναβλήθηκε. Δεν ξέρω πότε θα το εμβάλουμε στην ημερήσια διάταξη. Πρέπει όμως, γιατί η αναβολή έγινε για να πάρουμε τις πληροφορίες της αντιπροσωπείας. Τώρα τις έχουμε. Και πλέον μπορούμε να βάλουμε πάλι την έκθεσή σας στην ημερήσια διάταξη. Ωραία. Συνάδελφοι, προτείνω να καταλήξουμε τώρα κάπου. Ξέρω και κατανοώ ότι μπορεί να υπάρχουν ε, πληθώρα πληροφορίες και πολλές πιέσεις επίσης. Έτσι όπως καταλαβαίνω εγώ την κατάσταση και όπως είπε και ο συνάδελφος Μαρινέσκου που πήγε πριν από 1,5 χρόνο στην Ιγναλίνα και αν βέβαια αντιλαμβανόμεθα ότι υπάρχει πρόοδος το είπε η Κομισιόν και είναι σημαντικό αλλά βραδία υπερβολικά βραδεία. Και γι' αυτό πήγε η αντιπροσωπεία. Γιατί υπήρχε ειδική έκθεση από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. Αυτό έπρεπε να το λάβουμε υπόψη. Πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε τι μήνυμα θα στείλουμε σε όλους τους συμμετέχοντες και τους εμπλεκομένους. Όπως λέμε στα συμπεράσματά μας, νομίζω ότι θα πρέπει ως Κοινοβούλιο να αποστείλουμε στεναρό μήνυμα. Θέλουμε επιτάχυνση. Θέλουμε για την πυρηνική ασφάλεια και προς το συμφέρον των πολιτών θέλουμε να επιταχυνθεί όλο το πρόγραμμα και αυτό είναι ένα σαφές μήνυμα. Και αυτό είναι και ένα πόρισμα της αντιπροσωπείας που μπορούμε να κρατήσουμε. Νομίζω ότι καλό είναι να μείνουμε στο κείμενο που έχουμε. Δύο σχόλια για να απαντήσω στον συνάδελφο Μαρινέσκου. με κάπως από τη δήλωσή του ότι η συνθήκη προσχώρησης είναι αφηρημένη και έχει γενικόλογη διατύπωση. Δεν συμφωνώ, δεν μπορώ να συμφωνήσω με αυτή τη δήλωση ότι η, η συμφωνία προσχώρησης ε, ε, περιλαμβάνει ασαφείς προϋποθέσεις σε σχέση με τις προϋποθέσεις και τους όρους ένταξης. Ευχαριστώ. Η κυρία Γκρέσλε. Πρώτον, εδώ κάνει πάρα πολύ κρύο. Δεύτερον, ε, ε, Σιγμάντας. Καταλαβαίνω, καταλαβαίνω ε, και πραγματικά και εγώ δεν θα ήξερα ε, τι να κάνω αν είχα από πίσω την κυβέρνησή μου να με πιέζει. Εμεί, εγώ καταλαβαίνω τη διαφορετική σου άποψη, αλλά λυπάμαι πολύ. Τι να κάνω. Κατέληξα σε διαφορετικό συμπέρασμα και άλλοι μαζί που ήταν. Δεν γίνεται, δεν μπορούμε. Όμως έδωσες μάχη γενναία. Και η κυβέρνηση που σε πιέζει τώρα πρέπει να στο ε, αναγνωρίσει αυτό. Ότι έδωσες γενναία μάχη. Αλλάζω λοιπόν τη λέξη frozen στο κείμενο, παγωμένη στη suspended, να ανασταλεί και πρέπει να σταματήσουμε εδώ και να αποστείλουμε σαφές μήνυμα σε όλους τους εμπλεκομένους. Και σας διαβεβαιώνω, διαβεβαιώ, κύριε Πρέσβη, και διαβεβαιώστε και τη λιθουανική κυβέρνηση ότι εύκολα θα πείσετε την Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμών αν, τα αποτελέσματα προχωρήσουν σωστά. Εάν σε δύο-τρία χρόνια ε, διαπιστώσουμε και εμεί και το ελεγκτικό συνέδριο βέβαια θα μας ε, το διαβεβαιώσει αυτό ότι έχουν λυθεί τα προβλήματα και έχει επιταχυνθεί η διαδικασία, νομίζω ότι ε, εύκολα θα πιστούν οι συνάδελφοι εδώ από όλα αυτά. Καλώς, ευχαριστώ. Τελειώσαμε την απογευματινή μας ημερήσια διάταξη. Ευχαριστώ πολύ όλους τους συμμετασχόντες στο τέλος της δημόσιας συνεδρίασης. Λοιπόν, κλείνουμε την δημόσια συνεδρίαση. Κύριε Μαρινέσκου, θα σας ενημερώσω σχετικά με το πότε θα βάλουμε στη ημερήσια διάταξη την έκθεσή σας. Ευχαριστώ την Κομισιόν, το Ελεκτικό Συνέδριο, τους συνεργάτες της Γραμματείας και την, τους διερμηνείς και μετά από ένα σύντομο διάλειμμα παρακαλώ να προχωρήσουμε στην κλειστή συνεδρίαση των συντονιστών. Σε, λίγα, σε 3-4 λεπτά δηλαδή θα, συνεχιστεί, θα αρχίσει η συνεδρίαση των συντονιστών. Ευχαριστώ.